καλωσορίσω και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Πολιτισμού που λαμβάνουν μέρος σε αυτή την ακρόαση, αλλά όλους ιδιαίτερος θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Γκέγγεν Κουίν, την υποψήφιο Επίτροπο για τα θέματα της έρευνας, καινοτομίας και επιστήμης. Δεν χρειάζεται να κάνω μακρά παρουσίαση. Ξέρετε ότι για αυτή την ε, ακρόαση έχουμε σαφείς κανόνες σε ό,τι αφορά τον χρόνο ερωτήσεων και παρακαλώ όλους τους συναδέλφους και φυσικά και την ε, υποψήφια επίτροπο να παραμείνουν στα όρια του χρόνου ώστε και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος του καταλόγου αγορητών να έχουν και αυτή την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους. Όπως ξέρετε, σε αυτή την ακρόαση έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σημαντικό θέμα, το θέμα της καινοτομίας, της έρευνας, της τεχνολογίας και ξέρετε όπως και εγώ ο ίδιος ότι στον τομέα αυτό πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει ακόμα σημαντικές προσπάθειες. Έχουμε λοιπόν ένα σημαντικό έργο ενώπιόν μας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε διαβάσει το βιογραφικό της ε, κυρίας ε, υποψηφίας Επιτρόπου και τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο το οποίο της έχει δοθεί. Καταρχήν θα δώσουμε στην ε, κυρία Κίγκαν Κουίν τη δυνατότητα να κάνει μια παρουσίαση το πολύ 10 λεπτών και στη συνέχεια όπως προβλέπει ο κατάλογος θα τεθούν τα ερωτήματα από την πλευρά των βουλευτών. Δεν θέλω να θυμώσετε, αλλά θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ αυστηρός με την χρήση του χρόνου αγόρευσης. Αυτό είναι ένα θέμα στοιχειώδες ισοδικίας έναντι των συναδέλφων. Λοιπόν, θα δώσω λοιπόν τον <clears throat> λόγο στην κυρία Γκέγγεν Κουίν και νομίζω <clears throat> ότι έχετε δυνατότητα να παρουσιάσετε τον εαυτό σας ενώπιον της Επιτροπής μας και να κάνετε τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις για 10 λεπτά το μάξιμο. Κύριε Πρόεδρε. Η δημοκρατία, ο διάλογος και το πνεύμα υπολογότητος είναι βασικά για μένα. Εγώ πιστεύω ότι με την ε, σημερινή μου παρουσία θέλω να τονίσω την ε, σημασία αυτών των αρχών και ελπίζω ότι θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Ω πολιτικό που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την Ευρώπη και είναι προσιλωμένη στη δημοκρατία και την κοινοβουλευτική δημοκρατία ιδιαίτερα, θα ήθελα να σα παρουσιάσω τι πεπιθήσει μου, την εμπειρία μου και το όραμά μου. Από τότε που για πρώτη φορά ξεκίνησα ήταν συνδεδεμένη πάντα με το να εργάζεται η Ιρλανδία στα πλαίσια τη Ευρώπη και να μεταμορφώνει η Ευρώπη τι καρδιέ και τι ψυχέ των Ιρλανδών. Στη μακρά ε, καριέρα μου, σαν υπουργό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η δυνατότητά τη να αλλάξει το πλαίσιο των ανεπίλητων, όπω φαινόταν προβλήματα, ήταν πάντα μια έμπνευση για μένα. Στην υπουργική μου εμπειρία, εργαζόμενη για την ταχεία μεταρρύθμιση τη Ιρλανδία, ώστε να γίνει μια ειρηνική και προοδευτική κοινωνία και μια οικονομία τη γνώση δημιουργική, ήταν η ε, καινοτόμο δύναμη Ευρώπη σαν ήμουν μακρόν μέλο του Ευρωπαϊκού ε, Ελεκτικού Συνεδρίου και έτσι έχω καλύτερη γνώση για το πώ δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω σε, σε περιόδου κρίσεω εμεί στη δημόσια ζωή έχουμε ένα δημόσιο καθήκον να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό το κοινοβούλιο είναι ζωντανό μάρτυρα του πώ η πολιτική φαντασία για να καινοτομεί, να συμφιλιώνει και να ξεπερνά οδηγεί σε αποτελέσματα. 50 χρόνια ειρηνική συνύπαρξη, μια ενιαία αγορά, το ευρώ, μια ειρηνική επανένωση μετά τον ε, ψυχρό πόλεμο είναι, ε, επανενώνει την ήπειρό μας. Η Ευρώπη μας ε, διαμορφώνει την αλλαγή. Στην καρδιά της Ευρώπης είναι η καινοτομία. Είναι μια ένωση της καινοτομίας. Η ολοκλήρωση, η ένωση είναι η καινοτομία. Αντιμετωπίζοντας την άνοδο προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αλλαγής του κλίματος και το δρόμο προς λιγότερες εκπομπές άνθρακος, για μια στιγμή θα πρέπει να δούμε τι έχουμε πετύχει. Αν εγκριθεί η θέση μου, θα συνεχίσω να υποστηρίζω τις δημοκρατικές, κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας χρειάζεται να μετακινηθούμε από μια δεκαετία συζητήσεω για την Ευρώπη σε μια δεκαετία υλοποίηση έργων τη Ευρωπαίου. Η μεταμορφωτική, η μεταρρυθμιστική, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Πρόεδρου Μπαρόσο, οι πολιτικέ τεχνικέ γραμμέ το επιβεβαιώνουν αυτό. Η νέο χαρτοφυλάκιο για την έρευνα, καινοτομία και επιστήμη επιβεβαιώνει ότι θέλει ο κ. Μπαρόσο να πετύχει αυτό. Θέλω να προωθήσω την καινοτομία και την επιστήμη και την έρευνα στο επίκεντρο τη Ευρωπαϊκή Πολιτική. Να το πετύχει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει μια πραγματικά καινοτόμα ένωση. Ένα πολιτισμό καινοτομία οδηγεί σε αλλαγή, διαχείριση τη αλλαγή και ανοιχτό τρόπο προσέγγιση τι κάνουμε. Μια καινοτόμω ένωση θα υποστηρίζει αγορέ που είναι ανοιχτέ σε καινούριου ερχόμενου και που δίνουν κίνητρα επενδύσεις για, για να δοθούν επενδύσει για έρευνα. Η έρευνα δοκιμάζει τα σύνορα εφαρμόζει τεχνογνωσία και δημιουργεί κοινά αποτελέσματα, δίνει αποτελέσματα. Το θέλουμε. Καινοτομία τι σημαίνει, να ξέρει κανεί πότε να ανταγωνίζεται και πότε να συνεργάζεται σε ένα πλαίσιο διεθνέ πάρα πολύ σκληρό. Η γνώση, η έρευνα και η επιστημονική αριστεία είναι ακρογωνίω λίθο τη καινοτομία. Στη νέα οικονομία η λεπτομερή γνώση θα αντικαταστήσει το, α, το πετρέλαιο, το μαζούτ σαν κινητήρια δύναμη τη οικονομία. Σαν ένα τμήμα του οράματο 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει πολλέ μεταρρυθμίσει που θα επιταχύνουν και την καινοτομία ε, και θα γίνεται καινοτομία από την έρευνα μέχρι την πώληση. Βασισμένη στην κληρονομιά του Γιάννη Ποτότσινγκ που ήταν εντυπωσιακή, ένα κοινό όραμα για έρευνα, καινοτομία και επιστήμη θα πρέπει τελικά να χαρτογραφηθεί και να πετύχουμε αποτελέσματα. Από τώρα και στο εξή θα πρέπει να ε, διαμορφώνουμε τι πολιτικέ μα σύμφωνα με τι προκλήσει. Αυτή, αυτές οι μεταρρυθμίσεις οι ευρωπαϊκές για την έρευνα και την καινοτομία έχουν δύο στρατηγικούς στόχους. Πρώτον, να δημιουργηθεί μια νέα αγορά για την καινοτομία και δεύτερον να ολοκληρωθεί ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας. Θα πρέπει να χατογραφήσουμε και να δούμε πού είναι τα φράγματα και οι διελήψει όσον αφορά την καινοτομία. Μια νέα αγορά για την καινοτομία θα μπορούσε να προετοιμαστεί και να υλοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα μέλη αυτή τη Επιτροπή ρυθμιστικές απαιτήσεις, ε, διπλώματα ευαισθητεχνίας, δημόσιες προμήθειες και προδιαγραφές θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Μαθαίνοντας από τις ε, επιτυχίες που χρηματοδοτήθηκαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κίνητρα για επενδύσεις και χρηματοδότηση των μέσων της αγοράς για νέα έργα θα πρέπει να εξεταστούν. Στον πυλώνα τη έρευνα, αν εγκριθώ σαν μέλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δημιουργήσω μια πολιτική, ένα πλαίσιο ε, έρευνα με τρει προτεραιότητε. Πρώτα απ' όλα, ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα, να ασχοληθούμε με τι μεγάλε προκλήσει που αντιμετωπίζει η κοινωνία και να δημιουργήσουμε ε, έναν πολιτισμό, μια νοοτροπία έρευνα και καινοτομία. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα, θα πρέπει να ε, καθορίσουμε τι τρει πρωτοβουλίε ERA για καριέρε έρευνα, νέο προγραμματισμό, υποδομέ, μεταφορά γνώση και διεθνή συνεργασία. Θα πρέπει να κάνουμε την πέπτη ελευθερία για την κινητικότητα των ερευνητών, γνώση και την τεχνολογία σε όλη την Ευρώπη μια πραγματικότητα. Οι ερευνητέ μα θα πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν και να εργάζονται σε άλλα κράτη-μέλη και να απολαμβάνουν πλήρω προστατευμένη κοινωνική ασφάλιση και συνταξιωτικά δικαιώματα. Γνωρίζουμε ότι το 3% που είναι στόχο τη Βαρκελόνη είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για να επιτευχθεί θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κλίμα για επενδύσεις στην έρευνα. Η σημασία της ενθάρρυνσης έρευνας που είναι στα σύνορα της γνώσης μέσω ενός ανεξαρτήτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ερευνών δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Θα πρέπει να αποφύγουμε επικάλυψη προσπαθειών και κατακαιρματισμό μέσω καλύτερων κοινών προγραμμάτων. Δεύτερον, θα πρέπει να θέσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας στο επίκεντρο του προγράμματός μας για την έρευνα. Οι κλιματολογικές αλλαγές είναι ο τομέας εκείνος όπου η έρευνα άλλαξε και τις καρδιές και τα μυαλά. Επόμενο που πρέπει να κάνουμε είναι η έρευνα να διερευνήσει πώ οι κλιματολογικέ αλλαγέ θα επηρεάσουν τι ζωέ των πολιτών μας. Όσον αφορά την ενέργεια, θα πρέπει να υλοποιήσουμε τη στρατηγική ενέργεια και τεχνολογία, το σχέδιο SET και να επενδύσουμε σε ένα ευρύ φάσμα λύσεων, ούτω ώστε να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες. Όσον αφορά την υγιή γύρανση, χρειαζόμαστε νέες ιατρικές προσεγγίσεις, ούτω ώστε να μεταμορφώσουμε την ποιότητα διαβίωση των ανθρώπων σε μια γεράσια κοινωνία. Θα πρέπει να επικοινωνούμε το κοινό για να βλέπουν ποια είναι τα ωφέλη από την έρευνα. Θα είναι σημαντικό η υποστηριχτή πολιτική. Και τρίτον, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ένα, νοοτροπία για καινοτόμα έρευνα. Η έρευνα, όταν τη χειριστούμε σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε απίστευτη καινοτομία. Χρειάζεται να επιταχύνουμε την καινοτόμα έρευνα μέσω υποστήριξη κοινών ε, τεχνολογικών πρωτοβουλειών και να ετοιμάσουμε τι ε, συνθήκε αγορά σε σχετικέ αγορέ το τόπο εργασία έρευνα θα πρέπει να εξελιχθεί, ούτω ώστε περισσότερε γυναίκε να μπορούν να συμμετάσχουν στι επιστήμε. Θα πρέπει επίση να ασχοληθούμε με την αυξανόμενη αποσύνδεση μεταξύ επιστήμη και κοινωνία. Η κοινωνία θα πρέπει να γνωρίζει και να αισθάνεται άνετα με την επιστήμη που ε, βασίζει την πρόοδό τη, τη λειτουργία τη και την επιβίωσή τη. Η επιστήμη πρέπει να ανήκει στην κοινωνία το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας, ε, το 7ο για το 2007-2013 είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα, το δημόσιο πρόγραμμα στον κόσμο. Μέσα σε μια νέα πολιτική έρευνα και καινοτομία, το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να ειδωθεί σαν ένα μέσο και όχι σαν ένα αυτοσκοπό. Εγώ είμαι πλήρω δεσμευμένη να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματο πλαισίου 7 η υποτιμασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στοχευμένο τρόπο είναι βασική μα μέρημνα που χρειάζεται συγκεκριμένε αποφασιστικέ προσπάθειε στο μέλλον. Η απλούστευση τη χρηματο... χρηματοδοτική και διοικητική διαδικασία για το πρόγραμμα πλαίσιο 7 είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Χρειάζεται σωστή χρήση ε, των πόρων, ανάλογη έλεγχη και επαγγελματική διαχείριση. Θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την απλούστευση χωρίς να υπονομεύουμε τον έλεγχο ή την ποιότητα της αξιολογήσεως. Για τις ζωτικές συνεργασίες ιδιωτικού δημόσιου τομέα θυμαίνει ότι χρειάζεται να έχουμε φιλικότερους κανόνες και συνθήκες που βοηθούν την καινοτομία. Το Κοινοβούλιο μπορεί να δραματίσει ένα κρίσιμο ρόλο εξασφαλίζοντας συμπεφωνημένη α, θεσμική συνεργασία και συμφωνία σε αυτά τα θέματα. Ένα κόσμο μηδενικού κινδύνου είναι ένα κόσμο μηδενική καινοτομία. Τέλο, θα πρέπει να δούμε πώ να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικούς πόρους από τα διεθνωτικά ταμεία. Η Ευρώπη μπήκε στο έτος στην εποχή της καινοτομίας. Μπορούμε ή να ακολουθούμε ή να ηγηθούμε. Η Ευρώπη είναι στην καλύτερη της θέση όταν εργάζεται προς το μέλλον. Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με αυτή την Επιτροπή μπορούμε να προχωρήσουμε. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Πρέπει να κάνουμε τη διαφορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλή αρχή γιατί κερδίσαμε και χρόνο. Με τη σειρά τώρα θα δίνω χρόνο ενός λεπτού για ερώτηση, δύο λεπτών για απάντηση και πρώτη θα ακούσουμε την κυρία Πλάτρελ Καστίγιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε κυρία Τζόζεν Κουίν. Θα ήθελα εξ ονόματο τη ομάδα μου, τη ε, ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, να σα καλωσορίσω στην Επιτροπή Βιομηχανία. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα προχωρήσω αμέσω στο ερώτημα. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική απόφαση να ενώσουμε την έρευνα με την καινοτομία και την επιστήμη. Έτσι, ο πρόεδρος Μπαρόσο τόνισε την προσοχή του για την καινοτομία, φέρνοντας την καινοτομία στην καρδιά της προόδου και της ανάπτυξης της Ευρώπης. Αλλά όταν γίνεται μια τέτοια πρόοδος, βλέπουμε ότι όλα αυτά βρίσκονται σε ένα χαρτοφυλάκιο, τα θέματα της πρόοδου, και σε, άλλα, σε άλλο χαρτοφυλάκιο όλα τα άλλα. Για όλα τα θέματα της ε, καινοτομίας έχουμε από τη μία πλευρά τη σύνδεση με τη βιομηχανία, από την άλλη πλευρά έχουμε τη σύνδεση με τον πολιτισμό. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή τη σύγκρουση μεταξύ της θεωρίας της καινοτομία και των εργαλείων της ε, καινοτομία. Η κυρία Γκέγεν Κουίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Αντεκαστήλιο. Ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όταν παρουσίασε τι πολιτικέ του κατευθυντήρες γραμμέ στο Κοινοβούλιο ο κ. Παρόσο έθεσε στο κέντρο τη πολιτική του για την επόμενη <clears throat> επιτροπή την έρευνα και την καινοτομία, την πρόθεσή του. Εάν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τι παγκόσμιε προκλήσει, αν θέλουμε να εξέλθει η Ευρώπη από την οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, τότε είναι απαραίτητο να υπάρξει καινοτομία. Έχουμε τεράστιο ταλέντο στην Ευρώπη από ερευνητική άποψη. Έχουμε πολύ <clears throat> σημαντική έρευνα που έχει επιτευχθεί στην Ευρώπη. Όλα αυτά όμως πρέπει να μεταφραστούν σε θέσεις απασχόλησης. Είμαστε όλοι πολιτικοί και εγώ θα σας μιλήσω σαν πολιτικός. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο είναι να μεταμορφώσουμε την έρευνα σε θέσεις απασχόλησης και σε καινοτομία. Εδώ και πολλά χρόνια οι νέοι ενθαρρυνόντουσαν να σπουδάζουν και να μπαίνουν σε, στο χώρο της χρηματοοικονομικής οικονομίας. Τώρα είναι νεκρή αυτή η πτυχή της οικονομίας, δεν υπάρχουν νέες θέσεις. Γι' αυτό τους λέω, ας πούμε στον χώρο τον ερευνητικό, ας πούμε στον επιστημονικό κόσμο και ας προωθήσουμε την καινοτομία. <clears throat> σε σχέση με το ρόλο μου έναντι των άλλων επιτρόπων. Φυσικά διατρέχει εγκάρσια καινοτομία πάρα πολλά χαρτοφυλάκια. Και όπως αποφασίστηκε από τον Πρόεδρο και από τους άλλους επιτρόπους, εγώ θα έχω τον γενικό ρόλο του να εφαρμοστεί η πολιτική αυτή καινοτομία. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνοι μου. Χρειάζομαι όλου σα, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλέ δυσκολίε. Χρειάζομαι του συναδέλφου μου, του υποψήφιου επιτρόπου, οι οποίοι καλύπτουν διάφορε πτυχέ <clears throat> καινοτομία. Είτε είναι η ψηφιακή οικονομία, είτε είναι το επιχειρήν, είτε είναι η απασχόληση. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε και μόνο με τη συνεργασία μα θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο τη καινοτομία. Ευχαριστώ. Συμπληρωματικό ερώτημα. Ίσως υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί άλλοι έχουν τον έλεγχο της θεωρίας και άλλοι έχουν τις αρμοδιότητες και τον προϋπολογισμό. Αυτό φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολο για να μπορέσει να επιτύχει κανείς το στόχο αυτό. Παραμένει εκρεμές λοιπόν το θέμα αυτό της συνεκτικότητας και φαντάζομαι ότι απαιτεί την επιζήτηση κάποιων λύσεων Αλλιώς μπορεί αυτή η κατανομή των χαρτοφυλακίων να τροχοπεδίσει και όχι να προωθήσει την ε, καινοτομία, την έρευνα και την ε, επιστήμη. Κυρία Γκέγεν Κουίν, συμφωνώ φυσικά ότι υπάρχει μια δυσκολία πάντα αυτό ήταν το πρώτο βήμα να συνενώσουμε την καινοτομία, την επιστήμη και την ερεύνα σε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο θα οδηγήσει πολιτικά τη διαδικασία αυτή. Πιστεύω πρέπει να το κάνουμε αυτό, να προωθήσουμε πολιτικά αυτές τις ενέργειες. Πρέπει όμως συγχρόνως να προωθήσουμε την ανάπτυξη συμπράξεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Επίσης, η διευκόλυνση κατανομής κινδύνου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να προωθηθεί περισσότερο και να καταλάβει και νέους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι κυραχοκοκαλιά της βιομηχανίας που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Και ξέρω ότι η Επιτροπή σας λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην καινοτομία. Η καινοτομία χρειάζεται μια στενή συνεργασία με όλους τους επιτρόπους και κάθε επίτροπος στους τομείς όπου υπάρχουν σημεία συμφόρησης, θα πρέπει να κάνουν ότι μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα σημεία συμφόρησης και να δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ των διαφόρων τομέων. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω, απλώς θα συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Ριέρα Μαδουρέα. Ευχαριστώ πολύ, <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γκέγγεν Κουίν. Και εγώ εξ ονόματος της ομάδας μου θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ μάλλον για την παρουσίασή σας. Συμφωνούμε όλοι ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι βασικοί συντελεστέ βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κεφαλαιώδη στη στρατηγική την οποία εμεί θέλουμε να θεσπίσουμε για την έξοδο από την χρηματοοικονομική κρίση. Υπάρχει όμω μια άλλη πτυχή την οποία αναφέρατε και θέλω να υπογραμμίσω ότι από την έρευνα και την ε, καινοτομία θα πρέπει να βελτιώσουμε και την ποιότητα ζωής και την ευμάρεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό ήταν πάντα ο τελικός στόχος τουλάχιστον της δικής μου πολιτικής εργασίας. Πώς νομίζετε ότι η Κομισιόν μπορεί να συμβάλλει στο να προωθήσει και την κοινωνική διάσταση της έρευνας και της καινοτομία, ώστε πράγματι να εξυπηρετήσει τη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας, να βελτιώσει την παιδεία και την υγεία, τις συνθήκες εργασίας, την κοινωνική συνοχή, την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίας μέσα στην κοινωνία. Μέσα λοιπόν σε αυτό το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Χειροτομίας πώς μπορούν να προωθηθούν όλα αυτά. Απάντησε από την κυρία Γκίγκαν Κουίν. Ευχαριστώ. Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ε, είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι κάτι που αρχικά ξεκίνησε το 2000 ήταν μια μεγάλη ιδέα. Είπαν κάποιοι ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την προσπάθεια αυτή. Τι συνέβη. Λόγω τη συνθήκη τη Λισαβόνα και σαν Ιρλανδέζα ξέρω πολλά για τη συνθήκη τη Λισαβόνα σε αυτή τη φάση. Τι συνέβη λοιπόν. Το άρθρο 180 τη συνθήκη Λισαβόνα απαιτεί να δημιουργήσουμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα. Και το άρθρο 182 5, 5, μα δίνει τη δύναμη να κάνουμε, τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα. Από αυτό τον Ευρωπαϊκό Χώρο ε, έρευνας δημιουργήσαμε τα ευρωδίκτυα. Δηλαδή αφορούν το συντονισμό της έρευνας. Διότι γίνεται πολλή έρευνα στην Ευρώπη που είναι πάρα πολύ καλή, είναι άριστη. Στο τέλος όμως γίνεται σε διάφορες περιοχές και γινόταν πολλή επικάλυψη. Να σας ένα παράδειγμα. Στα Ευρωδίκτυο για τα ασφαλή τρόφιμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδε ότι υπήρχαν 72 διαφορετικές έρευνες που διεξήγονται ε, όσον αφορά το βακτηρίδιο της αλμονέδας. Είναι αλληλεπικάλυψη, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν σημαίνει συνεργασία ένωσης. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε και τις θέσεις απασχόλησης που θέλουμε για την οικονομία. Τι μπορεί να κάνει ιδιωτικό τομέα. Στο χώρο των ευρωπαϊκό της έρευνας, από το 2003, έχουμε αναπτύξει την Ευρω... τις ευρωπαϊκές βάσεις για τεχνολογία. Ε, ακολουθούν τη βιομηχανία, ξέρουν τι κάνει ο ιδιωτικό τομέα, ε, θέλουν να δημιουργήσουν θέσει απασχόλησης, 37 υπάρχουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν ευφυή δίκτυα, εξετάζουν θέματα ηλικής ενέργειας, δασοκομείας, όλους τους τομείς όπου υπάρχουν πιθανότητες δημιουργίας ε, θέσεων εργασίας για να βγούμε την οικονομική κρίση. Έχουμε αυτούς τους τομείς τις τεχνολογικές βάσεις. Και έτσι καταλήξαμε στις κοινέ τεχνολογικές ε, πρωτοβουλίες. Και ως μέλη της Επιτροπής ξέρετε ότι έχουμε πέντε από αυτές. Και έχω τη χαρά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, είχα τη χαρά να συναντηθώ, διακόπτει ο Πρόεδρος. Θα σας παρακαλέσω ε, να δώσουμε λίγο χρόνο και για τη, δευτε... για τη δευτερεύουσα ερώτηση, για τη συμπληρωματική ερώτηση της συναδέλφου. Ναι, κυρία Γκέγγεν Κουίν. Εγώ απλώς έθεσα αυτό το ερώτημα επειδή εφέτος είναι το έτος αγώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η Ισπανική Προεδρία είχε σχετικά προτείνει μέτρα για να ενισχύσει κοινωνικά μέτρα σε σχέση με την έρευνα και την καιροτομία. Τι εργαλεία και τι πρωτοβουλίες σκέφτεται να χρησιμοποιήσει προς την κατεύθυνση αυτή η Κομισιόν. Έχετε Παρακαλώ για να απαντήσετε. Καταρχάς, θα έπρεπε ασφαλώς να σημειώσω ότι η Ισπανική Προεδρία έχει ορίσει ως ε, κύριο τομέα προτεραιότητα στην ε, έρευνα. Έρευνα σημαίνει να εξετάζονται και όλοι οι τομείς που σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμεσα με την επίλυση και την αμείωση, την αντιμετώπιση της φτώχειας. Είτε πρόκειται για τα κράτη-μέλη, είτε πρόκειται για την, ε, τον υπόλοιπο κόσμο, θα πρέπει αυτό να το δούμε ως ένα πλέγμα. Ιδιαίτερα όμως πρέπει να προσφέρουμε λύσεις για τη μείωση της ε, φτώχειας, σε πολιτικές επιλογές και μόνο με πολιτικές επιλογές μπορούμε να τα καταφέρουμε πιστεύω, γιατί μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό και να ε, το αντιμετωπίσουμε, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε και μία ε, δράση αποφασιστική, να δρούμε εγκαίρως και να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Και εδώ χρειάζεται πολιτική βούληση. Ευχαριστώ, κυρία Εκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δική μου ερώτηση έχει να κάνει με δύο πτυχές το, της ερευνητικής πολιτικής. Την δέσμευση καταρχάς για συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και ε, δημόσιου τομέα στην έρευνα ιδιωτικών και δημόσιων ερευνητικών κέντρων, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μέχρι πρόσφατα 39% της συμμετοχής ε, στα ερευνητικά προγράμματα το προσέφερα ε, ο ιδιωτικό τομέα, ενώ τώρα έχει αυτό μειωθεί στο 25% λόγω της πολύ βαριάς γραφειοκρατίας που επικρατεί. Τι νομίζετε ότι θα μπορούσε ή θα έπρεπε να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και δεύτερον οι μεγάλες επιδημίες ή μάλλον οι μεγάλες αρρώστιες που ταλανίζουν τον άνθρωπο ε, και η δυνατότητα για τη μετώπιση τους χάρη στη χρήση της βιοτεχνολογίας και της έρευνας ε, στη βιοτεχνολογία. Σημαντικές ε, πτυχές των εφαρμογών της έρευνας είναι η έρευνα στα βλαστοκύτταρα. Ποια είναι η θέση σας απέναντι σε αυτήν την έρευνα. Απάντηση. Καταρχάς, το πώ θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Έχετε απόλυτο δίκιο και όταν μου έδωσε την, ε, το χαρτοφυλάκιο αυτό ο κύριο Μπαρόσο μου είπε ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να εξετάσω το θέμα τη απλούστευση. και ίσω γι' αυτό θεώρησε ότι είμαι καταλληλότερη για τον τομέα αυτόν. ακριβώ, διότι το ελεγκτικό συνέδριο ήταν το πρώτο θεσμικό όργανο το οποίο με δραστηριότητα ελεγκτική επεσήμανε ότι χρειάζεται να, υπάρχουν διαφορετικές, ε, να υπάρχει διαφορετική ένταση διαφορετικού τομεί τη ε, ευρωπαϊκή λειτουργία των ευρωπαϊκών οργανισμών. Και η απλούστευση ω προ τη γραφειοκρατία μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικού τρόπου που πρέπει να αναπτυχθούν. Αλλά βέβαια θα ήθελα να πω και σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα που έχουμε αυτή τη στιγμή ήδη εν λειτουργία, πώ ε, έχουν ήδη προχωρήσει. Σε ποιο βαθμό δηλαδή έχει προχωρήσει η απλούστευση ήδη από το 7ο πρόγραμμα. Έχει μειωθεί ο χρόνο αναμονή από τη στιγμή που υποβάλλεται μία πρόταση μέχρι την ώρα τη ε, έγκριση. Ε, για μέχρι ένα ορισμένο κόστο είναι πολύ πιο απλέ οι διαδικασίε. Κόστο προγράμματο ή σχεδίου. Υπάρχει μία μονοθυριδική δυνατότητα προσέγγισης για την εγγραφή, όταν υπάρχουν δηλαδή διαφορετικά προγράμματα ερευνικά, αντί να πρέπει τακτικά κανείς να καταθέτει τις ίδιες ε, πληροφορίες, έχει μία μονοθυριδική προσέγγιση και 15.000 άνθρωποι είναι ήδη καταγεγραμμένοι σε αυτό το σύστημα. Επίσης το ελεκτικό συνέδριο έχει κοιτάξει μια διαφορετική πτυχή, η οποία είναι πολύ σημαντική πιστεύω για την απλούστευση. Δηλαδή, είπε το ελεκτικό συνέδριο, στηριζόμενο σε κάποιο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα πρέπει να δούμε και ένα αποδεκτό ποσοστό σφάλματος, αποδεκτό μεν, το οποίο όμως δεν θα είναι ε, επιτρεπτό και να ανατρέπει τις βασικές αρχές της χρηστής διοίκησης. Αυτό ε, σημαίνει ταυτόχρονα ότι μπορούμε, μπορούμε να επιτύχουμε αυτή τη βελτίωση του ποσοστού σφάλματος και των ε, επιπτώσεων του κυρίως με λιγότερους κανόνες, με λιγότερη, με λιγότερη γραφειοκρατία. Γιατί λιγότεροι κανόνες σημαίνουν και λιγότερα σφάλματα και αυτό ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπήρχε μια δεύτερη ερώτηση. Ναι, αλλά θα ίσως η κυρία Εκ να σας δώσει την ευκαιρία με τη συμπληρωματική της ερώτηση. Κυρία Εκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ ναι, διαγνώσκω μια δέσμευση από πλευρά σας να, να αγωνιστείτε κατά της γραφειοκρατίας και να προωθήσετε την απλούστευση. Αλλά θα σας παρακαλέσω τώρα να ε, μου απαντήσετε στη δεύτερη ερώτηση, δηλαδή ποια είναι η θέση σας έναντι της ε, πολιτικής, τρέχουσας πολιτικής σας προς την αντιμετώπιση των μεγάλων, ε, των μεγάλων νοσημάτων που ταλανίζουν τον άνθρωπο, όπως το διαβήτη και άλλα. Απάντησε. Είναι πολλές οι ερευνητικές προσπάθειες που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή, ορισμένες των οποίων αναφέρονται στις ε, νευροεκφυλιστικές ε, νόσους όπως του Αλσχάιμερ. Και στόχος αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι να ε, εξασφαλίσουμε όχι μόνο περισσότερα χρόνια ζωής για τον άνθρωπο, αλλά και καλύτερα χρόνια ζωής πιο υγιή δηλαδή χρόνια ζωής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα και έρευνα την οποία θα μπορούν οι επιχειρήσεις, οι φαρμακευτικές ε, ε, να την αξιοποιήσουν έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη ζωή, περισσότερα χρόνια υγείας και να αντιμετωπίσουμε αρρώστιες όπως ο διαβήτης, η Αλσχάιμερς κτλ. Εν τέλει αυτό θα είναι το αποτέλεσμα και θα έχουμε διαθέσιμα για τους ε, πολίτες μας φάρμακα τα οποία θα βελτιώνουν τη ζωή τους. Και έτσι θα αλλάξει και η πολιτική της, των κυβερνήσεων. Ο κύριος, Μπουτικόφερ, κυρία Γκίγκεν Κουίν, θέλω να σας χαιρετήσω και να σας καλωσορίσω ιδιαίτερα ένθερμα από τους πράσινους και γι' αυτό, επειδή προέρχεστε από ένα πράσινο νησί, σας αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερα, ιδιαίτερη ευμένεια. Στα γραπτά, στις ε, απαντήσεις στα γραπτά ερωτήματα, και στην παρουσία σας δεν αναφέρατε καθόλου την έννοια της ανθρωποκεντρικής καινοτομία. Το όραμά σας για την καινοτομία και την ερευνητική πολιτική περιλαμβάνει μια τέτοια ανθρωποκεντρική σύλληψη της έρευνας και της καινοτομία. Γιατί αυτό σημαίνει κάτι περισσότερο από το να εστιάσουμε μονάχα στην καινοτομία σε επίπεδο προϊόντων. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια αντίληψη της πολιτικής καινοτομία που λαμβάνει υπόψη και τους στόχους του περιβάλλοντος και τους κοινωνικούς στόχους. Το ερώτημα είναι με ποιους ενδείκτες θα μπορούσατε εσείς να εκτιμήσετε την καθαρή κοινωνική προστιθέμενη αξία των πολιτικών καινοτομία μας και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την κοινωνική αξιοπιστία της πολιτικής καινοτομία. Κυρία Κουίν. Μα φυσικά η πολιτική καινοτομία θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα μεγάλα προβλήματα σε επίπεδο κοινωνία, τι μεγάλε προκλήσει που όλοι μα, σαν μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του κόσμου, πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ποιε είναι αυτέ οι προκλήσει. Καταρχήν, όπω είπατε, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η κλιματική αλλαγή. Αν δούμε έξω από τα, από τα παράθυρά μα, βλέπουμε τι γίνεται. Αυτό είναι ένα τομέα όπου η έρευνα έχει αλλάξει την ανθρώπινη νοοτροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το έχει επιτύχει η έρευνα. Η ενεργειακή απόδοση βασίζεται σε έρευνα, ε, εφαρμογή, καινοτομία μάλλον και εφιά εφαρμογή. Και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναθεωρηθεί εφέτος. Το πακέτο ανάκαμψης, το οποίο ανεκρίθηκε από την Κομισιόν το 2009, θέσπισε κοινοπραξίε δημόσιου ιδιωτικού τομέα, ιδίω στου τομεί που αναφέρατε. Πιο αποτελεσματικά ενεργειακά κτίρια, πράσινα αυτοκίνητα, εργοστάσια τα οποία είναι πιο οικολογικά. Όλα αυτά που μα επιτρέπουν να ζήσουμε σε ένα πλανήτη και σε ένα κλίμα με βιώσιμο και αηφόρο τρόπο, με χρήση <clears throat> ενεργειών οι οποίες θα μπορέσουν να είναι ανανεώσιμες και αηφόρες. Να μπορέσουμε λοιπόν να εμπλακούμε περισσότερο σε τομείς οι οποίοι είναι καθοριστικοί για το μέλλον μας <clears throat> και που θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο και πιο καθαρό περιβάλλον και ένα καθαρό πλανήτη όχι μόνο για εμάς αλλά και για τα παιδιά μας και τα εγγονιά μας και δυσέγγονά μας στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπιτεκόφερ, αν έχετε συμπληρωματικό ερώτημα. <clears throat> Χωρίς μικρόφωνο κύριε Μπιτεκόφερ. Η δυνατότητα πρόσβαση στα αποτελέσματα τη έρευνα. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο περιλάμβανε εν αυτή τη ενία και ε, την ιδέα ενός τορβανά της γνώσης. Σκοπεύεται λοιπόν να προαγάγεται αυτή την ιδέα, την ανταλλαγή δηλαδή ε, των γνώσεων που σχετίζονται με την, να την καινοτομία, να έχει κανείς τη δυνατότητα πρόσβασης και να μοιράζεται με τους άλλους γνώσεις. Βεβαίως, απάντησε, και ενθαρρύνω αυτή την ιδέα, αλλά για να υπάρξει η πρόσβαση στη γνώση που παράγουν οι ερευνητές Ευρώπης, πρέπει να εξασφαλίσουμε προηγουμένως μερικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη δική μου τη δουλειά, αλλά και με άλλους επιτρόπους. Σε παραδείγματι, πρέπει να κοιτάξουμε τα θέματα της πνευματικής διοκτησίας, εμπόδιο προς την κοινή χρήση της γνώσης. Πρέπει να δούμε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το κόστος κατοχήρωση ενός διπλωμάτος ευρεσιτεχνίας που είναι 20 φορές υψηλότερο από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Μεγάλη απόσταση βεβαίω έχουμε διανύσει τα τελευταία αυτά χρόνια, τα 20 αυτά χρόνια αν θέλετε, αλλά ε, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Και με τον κύριο Μπαρνιέ, εφόσον εγκριθούν οι υποψηφιότητε μα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σπεύω να συνεργαστώ στενά έτσι ώστε να κάνουμε ακόμη τα τελευταία αυτά απαραίτητα βήματα, έτσι ώστε οι διάφοροι φραγμοί στην προστασία τη πνευματική διοκτησία και τα διπλώμα, την κατοχήρωση διπλώματων ευρεσιτεχνία να αντιμετωπιστούν. Όπως είπα, πρόκειται για θέματα που δεν έχουν μόνο να κάνουν με το δικό μου τομέα αρμοδιοτήτων, αλλά με όλων των άλλων συναδέλφων τα χαρτοφυλάκια και θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι σκληρά για να διαφυλάξουμε αυτή την ε, εξαίσια γνώση που παράγεται στην Ευρώπη για να εξασφαλίσουμε ένα πλανήτη καλύτερο για μας και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας έτσι ώστε όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την έρευνα χωρίς κίνδυνο να την ε, ανατρέψουν, να την αναιρέσουν. Ευχαριστώ. Ο λόγο για ο κύριος Τσίσεστερ τώρα. Κυρία Γκέγκεν, τονίσατε στα σχόλιά σας τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Κάτι πολύ ευπρόσδεκτο. Όμως να τονίσω ότι από εσά περιμένουμε τις πρωτοβουλίες. Τονίσατε την εμπειρία σας στο ελεγκτικό συνέδριο για την μετώπιση του σημαντικού προβλήματος του διοικητικού άχθους που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές και αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Ρωτώ, θα είσαστε επίτροπος έρευνας που θα βρει την μεγάλη ιδέα, κάτι που έκανε προκάτοχή σας ή κάποιος που θα κάνει να λειτουργήσουν καλύτερα τα εφιστάμενα μέσα. Και κάνοντας αυτό, θα εφαρμόσετε, θα εξακολουθήσετε να εφαρμόζετε την αρχή της αριστείας Έχετε το λόγο, κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα είμαι πολιτικός και δεν είμαι δημόσια υπάλληλο. Αυτό είναι το πρώτο. Υπάρχει. Ε, ε, είπαμε πολλά, ήρθε η ώρα για δράση. Και θα ξεκολουθώ να μιλάω για την έρευνα και θα δώσω αποτελέσματα με την έρευνα που διαθέτουμε στους τομείς που χρειάζεται πολύ. Το δεύτερο είναι σωστό. Θα δώσω αποτελέσματα σε αυτήν την έρευνα. Θα χρησιμοποιήσω, όπως αποκαλύψατε σωστά, τα μέσα, κύριε Τσίστερ, τα εργαλεία τα οποία ήδη υπάρχουν, ούτω ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα στους τομείς που χρειάζεται η έρευνα για τη διόρθωση προβλημάτων και υπάρχουν πολλά προβλήματα στην κοινωνία που μπορούν να διορθωθούν να χρησιμοποιήσουμε την έρευνα που έχουμε. Όπως είπα, πολλοί γνωστοί είναι εδώ στα Κροατήριο, πολλοί θα με γνώριζαν ω πολιτικό στην Ιρλανδία και θα ξέρουν ότι είμαι ένα άνθρωπος των πράξεων. Δεν λέω ναι σε όλα, θα είμαι στεναρή όσον αφορά την προώθηση του προγράμματος αυτού. Δεν ασχολείστε με, δεν έχετε δημόσια υπάλληλο, λυπάμαι που το λέω αυτό. Εδώ έχετε μια πολιτικό απέναντί σας που θέλει δράση, θέλει πράγματα να γίνονται, θέλει αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τίτσεστερ, επερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν, ποια θα είναι η στάση σας έναντι κάποιων μεγάλων προγραμμάτων που έχουν ξεκινήσει. Σύνδεξη. Ίτερ. Fusion μάλλον, Ίτερ και Γαλιλαίος ε, που είναι σημαντικά προγράμματα ε, υψηλής τεχνολογίας που παίρνουν υποστήριξη ε, από τα διάφορα κονδύλια για τα ερευνητικά προγράμματα. Απάντηση. Τα κονδύλια για την έρευνα πρέπει να υποστηρίζουν και τα μεγάλα και τα μικρά προγράμματα. Θα μου πει τώρα ο Πρόεδρος ότι δεν έχω χρόνο. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα ITER ε, το πρόγραμμα το πειραματικό για θερμοπυρηνικούς αντιδραστήρες. Ε, είναι βασικό στοιχείο μακροπρόθεσμα στρατηγικής της Ένωσης για βιώσιμη, ε, βιώσιμο φοδιασμό ενέργειας. Δεν αφορά μόνο την Ένωση, βέβαια είναι διεθνές πρόγραμμα. Η Ένωση είναι ο οικοδεσπότης, αλλά έχουμε και άλλους εταίρους που συμμετέχουν εξίσου και πρέπει να του ενθαρρύνουμε. Είναι το μόνο πρόγραμμα, τολμώ να πω, που εξετάζει μια παγκόσμια πρόκληση για την καθαρή ενέργεια. Σημαντικό να παραμείνει. Όχι πάση θυσία όμως. Αυτό πρέπει να κάνω στο εγγύς μέλλον, αν επιβεβαιωθώ στη θέση μου, είναι να εξετάσω όλες τις πτυχές. Θα υποβληθεί έκθεση προόδου, θέλω να δω τι θα περιέχει. Υπάρχουν θέματα, θα ξέρετε και εσείς και η Επιτροπή, όσον αφορά τις εκτιμήσεις των δαπανών, και το ξεπέρασμα των ορίων του προπολογισμού. Μόλις έρθει η έκθεση θα κάτσω να τη δω. Χρειάζεται σωστή αποτελεσματική διαχείριση. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το μόνο πρόγραμμα που εμείς και οι διεθνείς μας, μας εταίροι ε, χωράει και λειτουργεί καλά και υποστηρίζεται. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εξ της ομάδας μου και εγώ θέλω να καλωσορίσω την κυρία υποψήφια Επίτροπο. Έχουμε μιλήσει πολύ εδώ για υποδείγματα έρευνας, για χρηματοδότηση και τρόπους για να επιτύχουμε την καινοτομία. Αλλά κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει πολύ πιο μεγάλο ποσοστό επισφαλών θέσεων για τους επιστήμονες στην Ευρώπη. Πολλοί λοιπόν έχουν πρόβλημα να μπορέσουν να επιτύχουν το στόχο αυτό να κάνουν την Ευρώπη μια, την πιο ανταγωνιστική κοινωνία του κόσμου. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση των επιστημόνων. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν θέσεις εργασίας. Αναρωτιέμαι αν αυτό μπορεί να είναι συμβατό με το όραμά σας και ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα λάβετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα το όλο και πιο μεγάλο των επισφαλών θέσεων εργασίας που πλήττει όλους του, πολλούς επιστήμονες σε ευρωπαϊκές χώρες. Σε διάφορε τομείς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκίγκον Κουίν. Το είπα και στην ενακτήριο δήλωσή μου. Την ελεύθερη κινητικότητα των ερευνητών με την εθαρρύνουμε. Και αν θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκό χώρο έρευνα που εξυπηρετεί το σκοπό μας, αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα που ενθαρρύνει τους ερευνητές να ενταχθούν στο σύστημα, να παραμείνουν στο σύστημα, να μπορούν να μετακινούνται και στα 27 κράτη-μέλη εύκολα, χωρίς να ανησυχούν για τις συνθήκες εργασίας τους, για τα συνταξιωτικά τους δικαιώματα, τα δικαιώματα τους κλπ. Και ένα από τα θέματα που ενδιαφέρει και το εξή ότι η Ισπανική Προεδρία απεφάσισε ένα κοινό διπουργικό συμβούλιο, στο οποίο δεν συμμετέχουν μόνο οι Υπουργοί Καινοτομία και Έρευνα, αλλά και οι Υπουργοί Απασχόληση, Υπουργοί Εργασία. Αυτό είναι πολύ καλή πρωτοβουλία, διότι πρέπει να συνεργαστούμε. Όπω και εγώ πρέπει να συνεργαστώ με τον συνάδελφό μου, ούτω ώστε οι συνθήκε εργασία που εμποδίζουν τη μετακίνηση την ελεύθερη των ερευνητών στα 27 κράτη μέλων, 67 ε, κράτη μέλη να αρθούν τα εμπόδια. Πρέπει να υπάρχουν κατά συνθήκε να τα κινούνται εύκολα. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε τον συνάδελφο για να πετύχουμε ακριβώς αυτό, ελεύθερη διακίνηση των ερευνητών. Κυρία Ματίας, για, για συμπληρωματική. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θέσω και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο. Υπάρχει μια τάση όλο και μεγαλύτερη για την συγκέντρωση των ερευνητικών πόρων υπάρχει στη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και αυτό είναι εύγλωτο. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη της κυρίας Επιτρόπου για το τι θα πρέπει να γίνει για να υπάρξει μια καλύτερη ενσωμάτωση των μικρών χωρών στην Ευρώπη στα συστήματα έρευνα και για να μπορέσουμε να καθορίσουμε καλύτερα ποιο είναι ο ρόλο των μικρότερων χωρών στο σύστημα έρευνα. Γιατί το σύστημα όπω το έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αρκετά άνισο και ει βάρο των μικρών χωρών. Ευχαριστώ, κυρία Γκίδεν είναι ένα από τα θέματα που μου έθεσαν αρκετοί συνομιλητές μου. Μέλη αυτής της Επιτροπής πριν από την ακρόασή μου. Αν δει κανείς και τα 27 κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαφορές πράγματι μεταξύ κρατών μελών. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να κάνουμε σίγουρα. Στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, τριτοβάθμια ιδρύματα για έρευνα, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ό,τι είναι αυτά, χρειάζεται εξυγχρονισμό. Στι μικρότερε χώρε χρειάζεται εξυγχρονισμό που φαίνεται δεν μπορούν να το πετύχουν όπω τα ήθελα. Δεν πρέπει να το κάνουμε όμω μόνο στο δικό μου τομέα, στο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρέπει να, δημιου... να κινητοποιήσουμε και διαθετικά ταμεία, να χρησιμοποιηθούν όπω χρησιμοποιήθηκαν στη δική μου χώρα για να δημιουργηθεί η οικονομία της γνώσης. Χρησιμοποιώντα λοιπόν πόρους από το πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά και τα 86 δις που είναι διαθέσιμα στα θετικά ταμεία να τα κινητοποιήσουμε. Ε, έτσι μπορούμε να κάνουμε πολύ χρήσιμα πράγματα. Να δημιουργήσουμε όχι μόνο υποδομές, αλλά και το δυναμικό που απαιτείται. Ακολουθεί η κυρία Τζαβέλα. Αγαπητή κυρία Γκέγγενγκάν, καλώς ορίσατε και εύχομαι όλα καλά για την, τον διορισμό σας. Καλή επιτυχία. Η ερώτησή μου ίσως είναι μια συνέχεια του κυρίου Τσίτσεστερ, αυτή τη στιγμή το θέμα της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς ή μη ειρηνικούς σκοπούς, προσέλεγχο δηλαδή, βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών σχέσεων. Ε, ας δούμε το Ιράν. Όμως εδώ και 10 με 15 χρόνια υπάρχει πλήρης έλλειψη επιστημονικού προσωπικού στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Πανεπιστήμια έχουν κλείσει τις παραγωγικές τους σχολές και είναι ελάχιστη η έρευνα που γίνεται στην πυρηνική ενέργεια. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για αυτό τον τομέα. Τι προτίθεστε να κάνετε εσείς ως καινούργια επίτροπος για να ενθαρρύνετε την πανεπιστημιακή έρευνα, την λειτουργία παραγωγικών σχολών μηχανικών στην πυρηνική ενέργεια ε, σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ κύριε Γκίγαν Κουίν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τζαβέλα. Συγγνώμη να δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Για την πυρηνική ενέργεια. Δεν υπάρχει μια χρυσή λύση, μια πανάκια που θα λύσει όλα τα προβλήματα της ενέργειας και του κλίματος. η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολείται και με την πυρηνική ενέργεια. Παραδείγματο χάρη το 7ο πρόγραμμα Ευρατόμ περιλαμβάνει αυτό και πτυχέ σχάση και σύνδεξη. Όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο μέρος της ε, έρευνας στη σύνδεξη είναι στα πλαίσια του προγράμματος ITER. Αλλά η πυρηνική ενέργεια παραμένει μια ε, τεχνολογία επιλογής σε πολλά κράτη-μέλη. Είναι μια, μια ενέργεια που δεν οδηγεί σε εκπομπή διοξίδου του άνθρωπου, Είναι μια τεχνολογία η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί σαν επιλογή των κρατών μελών που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την οδό. Είναι σημαντικό αυτό και είναι σημαντικό να το πω εγώ γιατί έρχομαι από μια χώρα που ξέρετε ποια είναι η πολιτική της. Η συνθήκη της Λισαβόνας τονίζει ότι το μείγμα ενεργειών είναι θέμα απόφασης κάθε μεμονωμένου κράτους. Και εμείς ως Κομισιόν δεν θα πρέπει να υπαγορεύσουμε ή να παρέμβουμε στα κράτη-μέλη να του πούμε τι είδους ενέργεια θα πρέπει να χρησιμοποιούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Δεν είναι η αρμοδιότητά μας ούτε ο ρόλος μας. Σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια παραμένει μια τεχνολογία που επιλέγουν ορισμένες χώρες και εάν με επικυρώσετε το διορισμό μου, εγώ θα διατηρήσω την έρευνα και την ανάπτυξή της για τις χώρες μέλες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια. Η κυρία Τζαβέλα για συμπληρωματικό ερώτημα. No more questions. Thanks. Thank you. Thanks very much. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Σωσαβάκνα, ο κύριος Σωσαβάκνα, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την κυρία υποψήφια επίτροπο, διότι προτάθηκε για αυτό το τόσο σημαντικό αξίωμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο προβλέπετε μέσα στο επόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο ανάπτυξης και έρευνα, να ενισχύσετε του οικονομικού πόρους για τους τομείς αυτούς ε, έρευνας που δεν συνδέονται άμεσα με την οικονομική κερδοφορία ούτε με τον χώρο του επιχειρήν. Δηλαδή, να ευνοήσετε την ε, έρευνα αυτή που μπορούμε ίσως προκλητικά να πούμε ότι δεν είναι αποδοτική οικονομικά, γιατί πολλές φορές <clears throat> η μη άμεσα αποδοτική έρευνα είναι αυτή η οποία σε μακροχρόνιο επίπεδο είναι και η πιο χρήσιμη. Αν φανταστείτε παραγωγός αν ο Καντ, το φιλοσοφικό του έργο θα μπορούσε να έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γκίγκαν Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ό,τι είδου έρευνα και αν είναι πάντα είναι αξιόλογη, χρήσιμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εξαρτάται από τη βιομηχανία, από τις ε, κυβερνήσεις, από τις εταιρικέ σχέσεις, τα διάφορα σχήματα που χρησιμοποιήσουν τη διαθέσιμη έρευνα. Υποστηρίζουμε το πρόγραμμα πλαίσιο που έχουμε για την έρευνα. Είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα με δημόσια χρήματα τον κόσμο. Και εντό αυτού ε, περιέχονται διάφορα, διάφορες έρευνες που στηρίζονται και στα 27 κράτη-μέλη. Όπως ξέρετε, σε ένα δίμηνο περίπου, θα γίνει ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου 7. Αυτή η ενδιάμεση αξιολόγηση θα εξετάσει όλους τους τομείς που συμπλαμβάνονται στο πρόγραμμα πλαισίου 7, όλες τις ερευνητικές πτυχές του προγράμματος πλαισίου 7 και τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως θα δείξουν που υπάρχουν προβλήματα, δυσκολίες, σε ποιους τομείς, που πρέπει να βοηθήσουμε, που υπάρχουν τομείς όπου χρειάζεται να σταματήσουν κάποια μέτρα. Θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τα αποτελέσματα. Θα τα εξετάσω εγώ τα αποτελέσματα τη διάμεση αξιολόγηση, να δω αν χρειάζεται να γίνουν αλλαγέ αμέσω στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνα και να εξετάσουμε και το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Τι χρειάζεται να αλλάξει ε, που πρέπει να είμαστε ευαισθηροί, τι πρέπει να προωθήσουμε με αποφασιστικό τρόπο από αυτά που είναι τώρα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Εστέ σίγουροι, δεν θα λησμονηθεί καμία έρευνα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Χρειάζεται όμω η ενδιάμεση αυτή αξιολόγηση να δούμε τι μα λέει, τι χρειάζεται να διορθωθεί. Και ό,τι χρειάζεται να διορθωθεί, εστέ σίγουροι ότι θα το διορθώσουμε. Συμπληρωματικό. Όχι, δεν έχω να θέσω άλλο ερώτημα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Όλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και συγχαρητήρια, αγαπητή κύριε μου, για το δυναμισμό, την αποφασιστικότητα που επιδεικνύεται. Θα έχετε 9 δισεκατομμύρια προπολογισμό. Όχι πολλά. Δεδομένων των προκλήσεων που έχετε απέναντί σα. Πώς διαβλέπετε την διαπραγμάτευση για τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές το 2013. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πολλά γίνονται σε επίπεδο κρατών μελών. Ήδη. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε η πολιτική της έρευνας να κοινοτικοποιηθεί και ως προς τη χρηματοδότησή της εσείς που ξέρετε πόσο ισχυρή είναι ε, οι εθνικοί εγωισμοί, ε, ίσως έχετε να μας πείτε μερικά πράγματα για το πώς θα μπορούσαμε σε κοινοτικό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες αυτές προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκενκουίν. Βεβαίω και θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί προετοιμαζόμενοι για αυτή την ε, ακρόαση έμαθα ότι με την διαφοροποίηση, τον κατακαιρματισμό της έρευνας χάνουμε πολλά από τα καλά αποτελέσματα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Άρα πρέπει ο ευρωπαϊκός χώρος της έρευνας να είναι ενωπιστικός να, να αντιμετωπιστεί κατά ενωτικό τρόπο έτσι ώστε να μην χάνεται, να μην κατακαιρματίζεται το αποτέλεσμα τη έρευνα. Χωρί να θέλω βέβαια εγώ να δίνω οδηγίε στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να κάνουν, αλλά με συντονισμό, με θέσπιση ενό ευρωπαϊκού χώρου έρευνα, πιστεύω θα έχουμε μια τεράστια ευκαιρία τον συντονισμό αυτόν να τον αναπτύξουμε για να μην υπάρχει επανάληψη, επικάλυψη της ίδιας έρευνας και βεβαίω είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, και για τι χρηματοοικονομικέ συζητήσει, για το διάλογο για τι μεσονομικέ προοπτικέ που θα έχουμε μπροστά μα. Και ασφαλώ Δεν θα σας ε, ξαφνιάσω αν σας πω ότι όταν πάει κανείς να στήσει χρήματα, είτε είναι επίτροπος, είτε είναι υπουργό, είτε είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν έρχεται η ώρα να μιλήσει λοιπόν για προϋπολογισμό, είναι μόνος του ε, και ε, έχει πολύ δύσκολο έργο να διεκδικήσει προ τώρα χρήματα. Αλλά είναι μια πρόκληση την οποία είμαι διατεθειμένη να αναλάβω. Το έχω κάνει και πριν από το θόκο τον ε, υπουργικό που είχα. Είμαι διατεθειμένη να το επαναλάβω και τώρα αυτό το εγχείρημα ω επίτροπο. Και επιπλέον η Επιτροπή είναι ένα συλλογικό όργανο. Καθένα αγωνίστε για το δικό του τομέα αρμοδιοτήτων και όταν μοιραστεί η πίτα αποφασίζει η Επιτροπή λίγο πολύ το τι μερίδο θα λάβει ο καθένα στο κάθε χαρτοφυλάκιο. νομίζω ότι θα, θα αγωνιστούμε για να έχουμε στο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Συμπληρωματική ερώτηση. Εάν έχετε ανησυχίε προ το Συμβούλιο, μπορείτε να στηριχθείτε στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου, γιατί θα είμαστε στο πλευρό σα. Και κυρία Επίτροπε, με συγχωρείτε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε, θα ήθελα να σα ρωτήσω εάν είστε διατεθειμένοι μαζί με τους συναδέλφους σας να θέσετε ένα τέρμα στα προβλήματα ελέγχου των ερευνητικών κονδυλίων, γιατί οι ερευνητές ε, βρίσκονται σε απόγνωση και λόγω των περίπλοκων κανόνων, αλλά και λόγω των ε, περίπλοκων και μη σύμφωνων με τους διεθνείς κανόνες λογιστικών ελέγχων ε, ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που τους φέρνουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είστε διεθυμένοι να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Απάντηση. Για, τους, για τον ιδιότερο ερευνητή και για τις μικρόμεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερως ερευνητικές επιχειρήσεις ε, που έχουν αναπτύξει δραστηριότητε με τα βάση τα προγράμματα αυτά και από τις τελευταίες εβδομάδες με την επαφή που είχα μαζί μου ακούω ότι βρίσκονται σε απόγνωση, ότι βρίσκονται στα όρια ε, της λογικής ως προς τις δημοσιονομικές, ε, προς τους ε, δημοσιονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν. Και αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι δεν θέλω εγώ να αναλάβω καμιά πρωτοβουλία ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να θέσει ένα αμφιβόλο την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Γιατί έχουμε να κάνουμε τα λεφτά του Ευρωπαίου Φορολογούμενου, έχουμε την υποχρέωση να τα σεβαστούμε και να τα χειριστούμε με τρόπο ορθό. Όμως, όπως είπα και σε άλλη περίσταση, νομίζω υπάρχουν τρόποι να απλουστεύσουμε τα πράγματα. Υπάρχει στρατηγική για, τα ενιαία, για, την, για τον ενιαίο λογιστικό έλεγχο που ήδη έχουμε πει ότι θα πρέπει να βρούμε διαφορετικούς τρόπους ώστε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικούς τομείς χάραξης πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, θέλει να προβάλλει την έννοια του αποδεκτού περιθωρίου σφάλματος με το σχετικό έγγραφο εφέτος και πάλι να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το σφάλμα αυτό, το, το ποσοστό αυτό σφάλματος και νομίζω ότι πάλι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε και ιδιαίτερα με εσά και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού που συμμετέχετε αλλά και από την Επιτροπή της ε, Βιομηχανίας νομίζω μπορούμε να βρούμε λύση. Αυτές οι δύο επιτροπές από κοινού μπορούν να βρουν τη σωστή λύση και να πείσουν ε, τον κόσμο ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και να εξετάσουμε τη δυνατότητα για ένα αποδεκτό ποσοστό σφάλματος και να αναπτύξουμε μια πολιτική η οποία είναι σωστή και η οποία δεν μπορεί να είναι και unisex. Πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές λύσεις και διαφορετικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τχοτμάν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Κίκεν Κουίν, είπατε ότι είστε πολιτικός. Το μήνυμα το λάβαμε. Πολιτική ερώτηση λοιπόν θα σας υποβάλω. Διαπιστώνουμε από την τωρινή κατάσταση ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι τη Λισαβόνα. Οι ερευνητές μας μας λένε ότι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και οικονομική και κοινωνική ε, έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στον τομέα αυτών, στην οικονομική, τα οικονομικά δεδομένα, στην οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την σημασία της γνώσης και της προστασίας ε, της γνώσης. Αυτός ο πυλώνας ε, του ευρωπαϊκού ε, χώρου που είναι το, 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, πώς θα μπορέσει να διαφυλαχθεί όταν βλέπουμε ότι ορισμένε χώρες μέσα από τη διαδικασία της Λουμπλιάνα είναι, είναι διατεθειμένες και προτιμούν από ό,τι φαίνεται να κάνουν έρευνα à la carte και πώς θα επιτρέψετε τη συνεργασία και με τα πανεπιστήμια, τα οποία, πράγμα το οποίο σημαίνει μερικές φορές αντιπαράθεση με τους ε, εθνικούς υπουργούς. Κύριε Κίγαν Κουίν. Θα είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να κερδίσουμε τους ερευνητές. Ξέρω ότι μερικές φορές θα βρεθούμε, όπως είπατε και εσείς, σε αντιπαράθεση με τα κράτη-μέλη, που ίσως να είναι αναγκαία, χωρίς να την προτιμώ βέβαια. Αλλά ίσως χρειάζεται και ο καθένας θα πρέπει να διαφυλάξει ε, και να αγωνιστεί για τα εφοετάχθη. Γι' αυτό λοιπόν όταν ένα επίτροπο έχει αναλάβει κάποιο χαρτοφυλάκιο, θα πρέπει να αγωνιστεί με βάση τα πιστεύω του, με βάση τα καθήκοντα που έχει αναλάβει. σω κάποια κράτη-μέλη να μην είναι ικανοποιημένα, κάποια άλλο, άλλα όμω θα είναι. Και θα πρέπει να στηρίξουμε του ερευνητέ για να επιτυγχάνουν του στόχου που ορίζονται για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία. Αυτό μπορούμε σε διάφορου τομεί. Δεν πρόκειται για την απλούστευση, δεν πρόκειται για τον ε, έλεγχο, εμπιστοσύνη και έλεγχο, για την οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, είτε πρόκειται για την ε, ε, ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προγράμματος ανάκτησης, ανάκαμψης με χρήση και ιδιωτικών και ε, δημόσιων πόρων. Να έχουμε δηλαδή μια βάση, μια ερευνητική βάση, μια βασική έρευνα η οποία θα έχει εφαρμογές και η οποία με την γεροτομία θα μας βοηθάει να προχωρήσουμε. αυτά με μια πολιτική καινοτομία που όπως είπα νωρίτερα δεν θα αναλάβω να συντάξω να διατυπώσω μόνη μου αλλά ολόκληρη η Επιτροπή και όλη η Επιτροπή μαζί και η δυνατότητα για συνεργασία, για συντονισμό ε, τη δουλειά που κάνουμε στα 27 κράτη-μέλη σημαίνει ότι μπορούμε να επιτύχουμε μια οικονομία της γνώσης που θα μας στηρίξει στο μέλλον, που θα μας προσφέρει μια καλύτερη κοινωνία για όλους, που θα μας προσφέρει τις θέσεις εργασίας που χρειαζόμαστε τόσο ε, γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε και να βγούμε από αυτή την οικονομική κρίση. Κυρία Τροτσμάν, για συμπληρωματική ερώτηση. Εφόσον πρόκειται για ερευνητέ, μπορώ να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι σας <clears throat> και επακριβώς μπορείτε να ποσοτικοποιήσετε τους στόχους σας σε ό,τι αφορά το ποσοστό γυναικών μεταξύ των ερευνητών. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα στην επιστήμη, η παρουσία των γυναικών. Σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας είναι σημαντικό αυτό, αλλά εγώ θα περιοριστώ στο θέμα της επιστήμης. Εγώ έχω κοιτάξει ποια είναι η θέση των γυναικών στην επιστήμη. Ξεκινούν να υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε. Μετά όμω κάνουν οικογένεια, υπάρχει πίεση από την οικογένεια, πρέπει να αποσυρθούν από τον ερευνητικό χώρο και μετά φαίνεται ότι είναι απίστευτα δύσκολο να επανέλθουν στον χώρο εργασία αυτό το οποίο θέλω να κάνω, να ενθαρρύνω περισσότερες γυναίκες <clears throat> να παραμείνουν στο χώρο της εργασίας και όταν σε, λίγες, ε, σε, προ, σε λίγη καιρό θα έχουμε στη, στο Δουβλίνο μια έκθεση για τους νέους, τα νέα παιδιά, να μπορέσουμε να τους πείσουμε να ενδιαφερθούν για το τομέα της επιστήμης και να αναζητήσουν εκεί θέσεις εργασίες εκεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια συναρμογή των συνδικών εργασίας και διαβίωσης και θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους βιομηχανικούς χώρους όπου οι γυναίκες έχουν καταφέρει να παραμείνουν στην, ε, στον τομέα της έρευνας και να πάρουν τα διδάγματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους κλάδους που δεν ήταν τόσο επιτυχείς από αυτή την άποψη. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό θέμα για μένα σαν γυναίκα που έχω παίξει, ελπίζω, ένα πρωτοπόρο ρόλο σε όλα αυτά τα θέματα. Δεν πιστεύω στις ποσοστώσεις, αλλά πιστεύω στους στόχους. Γιατί νομίζω ότι αν θέτουμε στόχους μπορούμε τότε να επιτύχουμε αποτελέσματα και μπορούμε να ελέγχουμε κατά πόσον επιτυχάνονται αυτοί οι στόχοι ή όχι. Η κυρία Νίμπλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Γιγκαν Κιν, Κουίν, <clears throat> εδώ είμαι από την άλλη μεριά. Εδώ, εδώ. Κυρία Γίγκαν Κουίν, θέλω να αναφερθώ και πάλι στο θέμα της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών. Υπήρξατε μέλος του ελεκτικού συνεδρίου και επομένως ο κύριος, το κύριο έργο σας ήταν να ελέγχετε τα, τα άλλα θεσμικά όργανα. Τώρα δεν είσαστε επίτροπος δημοσιονομικού ελέγχου, αλλά επίτροπος για τα θέματα έρευνας και κοινοτομίας. Ε, εγώ εδώ και 10 χρόνια που είμαι σε επαφή με τους εκπροσώπους του ερευνητικού κόσμου ακούω πάντα τα ίδια πράγματα, ότι υπάρχει μια τεράστια γραφειοκρατία που διέπει όλα τα προγράμματα έρευνας. Εσείς είστε, έχετε μια εμπειρία ως ελεγκτής λογαριασμών. Έχετε τη δυνατότητα να περάσετε από μια ε, αντίληψη που βασίζεται σε αποδείξεις σε μια ε, διαδικασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη προς τους ε, επιστήμονες. Τι καινούριο λοιπόν μπορεί να υπάρξει για να υπάρξει πραγματική διευκόλυνση και απλοποίηση των διαδικασιών. Τι έχετε να προτείνετε για όλα αυτά τα θέματα. Κυρία Γκίγαν Κουίν. Σας ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ. Η απλούστευση όπως σας είπα έκανα ένα σχόλιο προς τον κύριο Οντί. Το ελεκτικό συνέδριο, αν δει κανείς την απάντηση όσον αφορά αυτό το νέο ελέγχο, ήταν το πρώτο που δημοσίασε ένα έγγραφο αναφέρθηκε σε διάφορα ποσοστά σφαλμάτων σε διαφορετικούς ε, ε, τομείς πολιτικής και τη χρηματοδότηση αυτών. Και εξετάζουμε και το ανεκτό, το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου και θα εκδώσουμε σχετικά έγγραφο. Θα, εγώ θα υποβάλω ανακοίνωση, αν γίνω επίτροπος για επιστήμες, καινοτομία και έρευνα, θα υποβάλω ανακοίνωση αρκετά πρωί όσον αφορά την απλούστευση. Και Νομίζω ότι αυτή η διοργανική συζήτηση έχει ξεκινήσει όσον αφορά το κοινό αποδεκτό κίνδυνο, το κοινό αποδεκτό επίπεδο κίνδυνου. Θα, ε, αν γίνει αυτό θα μας υποστηρίξει και σας και εμένα αυτό που θέλουμε να κάνουμε και αυτό που θέλει να κάνει και η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού από αυτά που λέει και ο Σοντή. Όπω ανέφερα και με επιθυμήσατε, ανέφερα διάφορα πράγματα που είχα κάνει όσον αφορά την προσπάθεια για απλούστευση. Επίση, υπάρχουν και συμπληρωματικά πράγματα πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι θα ιδωθούν από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η ενδιάμεση ε, αξιολόγηση του προγράμματος Πλαισίου 7. Θα δούμε πού απομένουν περιοχές που χρειάζεται απλούστευση και πού όχι. Εγώ ακολουθώ μια απλή φιλοσοφία. Αν έχουμε λιγότερους κανόνες, έχουμε λιγότερα σφάλματα. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, ναι, θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να έχουμε ομοδοποιημένα ποσά, ναι, θα πρέ... ποσά, ναι, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Θα το δούμε κατά την αξιολόγηση του εβδόμου προγράμματος προγράμματο πλαισίου. Ακολουθούμε σωστό δρόμο, όλοι μπορούμε να συνεργαστούμε και χρειάζομαι σίγουρα την υποστήριξή σα για να τα καταφέρω σε αυτή την διοργανική συζήτηση που διεξάγεται πράγματι στον τομέα τη ε, απλούστευση. Ευχαριστώ. Κυρία Νίμπλα, ναι, σα ευχαριστώ για την απάντησή σα που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι τα μικρά προγράμματα έρευνας τα οποία θέλετε να διατηρήσετε θα πρέπει να υπόκειται σε πιο απλουστευμένες διαδικασίες από ό,τι για τα μεγάλα προγράμματα τα οποία πρέπει να έχουν πιο ενδελεχή ε, μορφή ελέγχου. Τώρα για, την, ε, για τη βιομηχανία είπατε ότι υπάρχει η μια μείωση της συμμετοχής του, των βιομηχανικών κλάδων στον τομέα της ε, έρευνας, πώς θα τους δώσετε περισσότερα κίνητρα για να επανέλθουν σε αυτό το χώρο, κύριε υποψήφια Επίτροπος. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε κίνητρα στη βιομηχανία, είτε είναι μισο, μικρομεσαία επιχείρηση, είτε είναι μεγάλη επιχείρηση που βλέπει σε παγκόσμιο επίπεδο προβλήματα. Αν είναι οι πρωτοβουλίες, ε, κοινέ πρωτοβουλίε ε, τεχνολογίε που πήγαν πάρα πολύ καλά, έχουμε πέντε από αυτές, Έχουμε μία που εξετάζει τα καινοτόμα φάρμακα που ασχολείται με αυτό το θέμα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ζωτικά. Έχουμε την πρωτοβουλία τη καθαρού εθέρε ε, που ενδιαφέρει πολύ τη βιομηχανία. Ε, θέλουμε να δούμε τη νέα γενιά αεροσκαφών. Ε, έχουμε κάτι για τις κυψέλες καυσίμων που αντικαθιστούν τη βενζίνη στα οχήματα. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες προέρχονται από τις τεχνολογικές βάσεις που έχουμε δημιουργήσει, που είναι ένας δρόμος που ακολουθούμε, ώστε η βιομηχανία εν γέννη, είτε οι μεγάλε επιχειρήσει, τα μικρομεσαίε επιχειρήσει να μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πλαίσιο, να μπορέσουν να συμμετάσχουν και να χρησιμοποιήσουν την έρευνα. Βέβαια, πολλές εταιρείε τώρα εξωτερικεύουν τι ε, ερευνητικές τους ανάγκες, Απευθύνονται αλλού, δεν κάνουν την έρευνα εντός της εταιρεία. Αναθέτουν εκτός την έρευνα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τώρα που είναι δύσκολα τα οικονομικά πράγματα, να ενθαρρύνουμε να τα κάνουν μόνες τους. Να δούμε τι έκανε η Φιλανδία. Αποφάσισε ότι η επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία ήταν η σωστή λύση για να αντιμετωπιστεί η κρίση που περνούσε η Φιλανδία τότε. Τώρα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να το κάνουν αυτό. Είναι μια τεχνολογία της γνώσης. Μιλάμε για τεχνολογία, για επένδυση για το μέλλον. Θέλουμε έρευνα που θα πηγαίνει μέχρι τον πολιτή, τον λιανοπολιτή. Θα πρέπει η έρευνα να χρησιμοποιείται ε, με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει αποτελέσματα. Ο κύριος Γκέρεκ. Κυρία Κουίν, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή: Μια αποτελεσματική εφαρμογή τη πανεπιστημιακή έρευνα εξαρτάται στο κατά πόσο μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και αντιμετώπιση του υψηλού κόστου που συνεπάγεται η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχει υψηλό κόστο όσον αφορά την προσβασιμότητα σε, νέα, σε νέε άδειε ευρεσιτεχνία και υπάρχει μακρά περίοδο προστασία και υπάρχουν και θέματα όσον αφορά το λογισμικό. Καθώ και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και φαρμακευτικά προϊόντα. Εξού και ερώτησή μου, ποιο είναι το πολιτικό σας όραμα το οποίο θα οδηγούσε σε μια ταχεία λύση όλων αυτών των προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα του, του πνευματική πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπος. Απάντηση. Κύριε Γκέρεκ, προηγουμένω αναφέρθηκα στο θέμα των διπλωμάτων ευσυτεχνία, την πνευματική ιδιοκτησία, που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Δημιουργεί προβλήματα, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε προχωρήσει πολύ σε 30 χρόνια, αλλά δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Έχουμε κάποιο δρόμο ακόμα που πρέπει να καλυφθεί. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι κάτι που αφορά και τον συνάδελφό μου τον κύριο Μπαρνιέ. Δεσμεύομαι απέναντί σα ότι θα συνεργαστώ στενά με τον κύριο Μπαρνιέ, αν και οι δυο μα εγκριθούμε, ούτω ώστε το τελικό βήμα να γίνει σε αυτό το τομέα. Είναι τεράστια σημασία σε αυτό για του ερευνητέ. Το κόστος χορηγήσεως διπλώματο ερευνητή στην Ευρώπη είναι 20 φορέ περισσότερο από ό,τι στη ΣΥΠΑ. Και ακόμα χειρότερα, για να διατηρηθεί μετά ίσως είναι 50 με 60 φορές πιο ακριβό από ότι είναι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Άρα θα πρέπει να βρεθεί ένας δρόμος για να ξεφύγουμε από αυτή την εμπλοκή, να ανοίξει ο δρόμος, να ανοίξει πόρτα, να δώσουμε την απαραίτητη προστασία και υποστήριξη που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι ερευνητέ και να είστε σίγουροι ότι εγώ θα ε, κάνω ό,τι μπορώ μαζί με τον κύριο Μπαρνιέ ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τα τελευταία βήματα που απαιτούνται σε αυτό το τομέα. Κύριος Γκέρεκ, κατά ερώτηση. Ε, ε, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Θα χρειαστεί πολύ θάρρος για να το αντιμετωπίσετε. Να πείσετε τους συναδέλφους σας ότι θα πρέπει και εκείνοι να το αντιμετωπίσουν, γιατί είναι όντως ακανθώδες. Απάντηση. Ελπίζω ότι η εμπειρία μου από την πολιτική μου σταδιοδρομία στην ε, Ιρλανδία θα, θα έχει αποδείξει ότι είμαι η θέση να ο θάρρος, τουλάχιστον από καιρούς καιρών. Όπως είπα, δεν είμαι από αυτούς που σκεύουν το κεφάλι, είμαι από αυτούς που παίρνουν αποφάσεις και που ε, προβαίνουν σε δράση. Έχουμε πολλά κάνει για την ε, ευρεσιτεχνία, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και θα τα κάνω μόνο μου. Θα συνεργαστώ στενά με τον κύριο Μπαρνιάν και εκείνος εγκριθεί στη θέση του ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα τελευταία εμπόδια, τους τελευταίους φραγμούς για την έρευνα στην Ευρώπη, ώστε εν τέλει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που να αντέχει η τσέπη του κοινού ερευνητή, που να μην τον φέρνει σε δυσμενή θέση σε σχέση ιδιαίτερα με τον ερευνητή από τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ κυρία Καμπάιο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε, όπως είπατε, ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας είναι θεμελιώδης για το μέλλον της Ευρώπης. Με ποιο τρόπο θέλει η Κομισιόν να προωθήσει τη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, κυρίω μέσα από τη σύνδεση των κοινοτικών προγραμμάτων με τα εθνικά προγράμματα χωρίς να χαθεί η, εθνική, η ευρωπαϊκή διάσταση. Αναφέρατε τα δίκτυα τα ευρωπαϊκά, αλλά αναφέρατε επίσης και το άρθρο 169. Πώς βλέπετε λοιπόν τη μελλοντική ανάπτυξη αυτών των εργαλείων και κατά πόσο θέλετε να δημιουργήσετε και νέα εργαλεία για να προωθήσετε τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Και πού βλέπετε τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας για να μπορέσει να συμπληρωθεί ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας. Ευχαριστώ. <clears throat> Κυρία Κουίν. Το Ερευνητικό Συμβούλιο δίνει το στοιχείο της αριστείας. Αυτό ήταν ο στόχος του, γι' αυτό πρέπει να έχει υποστήριξη και θα έχει τη δική μου υποστήριξη. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πρωτοβουλίες για να συμπληρώσουμε τον ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο που αναφέρατε κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες, μερικές είχα αναφέρει και εγώ ίδια, νομίζω ότι τα εργαλεία που έχουμε δεν επαρκή. Χρειαζόμαστε περαιτέρω εργαλεία περισσότερες πρωτοβουλίες. Χρειαζόμαστε και το άρθρο 169, έχουμε το μεγάλο πρόγραμμα bonus, το οποίο κοιτάζει την έρευνα σε όλη την περιοχή της Βαλτικής. Έχουμε το πρόγραμμα αντιμετώπισης του AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης, πάλι πρόγραμμα του άρθρου 169. Αυτά είναι δημόσια προγράμματα. Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά προγράμματα πάλι πρέπει να κινηθούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε τι κοινέ τεχνολογικέ πρωτοβουλίε που ανέφερα προηγουμένω, Είναι πολύ σημαντικέ για να δίνουν τη δυνατότητα να γίνεται έρευνα σε επίπεδο που θα αντιμετωπίσει τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές που αντιμετωπίζουμε όλοι ως Ευρωπαίοι. Χρειαζόμαστε να έχουμε και αγορές εχμής για τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι, παραγωγή χάρη, τα προστατευτικά ενδύματα για τους πυροσβέστες, για τους ψαράδες. Τα θέματα της ε, μετρήσιμης ενέργειας, η ηλεκτρονική η υγειονομική περίθαλψη, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία προχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πλατφόρμα μέσα από τις κοινέ πρωτοβουλίες και έχουν φτάσει σε αγορές οι οποίες είναι αγορές εχμής. Πρέπει να υπενθυμίσω επίσης ότι το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ένα σχέδιο ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εκεί υπάρχουν τρεις συμπράξεις, τα εργοστάσια του μέλλοντος, τα, η ενεργειακή απόδοση και τα πράσινα οχήματα. Μέσα λοιπόν από τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούμε να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο, μειώνοντας την αλληλοεπικάλυψη, επομένως την απώλεια ευκαιριών για τους Ευρωπαίους. Εάν προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική η οποία σε τελική ανάλυση θα δημιουργήσει θέσει εργασία. Αυτό είναι ο στόχο μα. κυρία Καρβάλιου, συμπληρωματικό ερώτημα. Θέλω να τονίσω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα μέσα στα πλαίσια τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα. Πώ θα μετατρέψει η κυρία Επίτροπο αυτό το Συμβούλιο για να μπορούν να συμμετέχουν και εθνικοί και περιφερειακοί φορεί και πώ θα εξασφαλίσει και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στο φορέα αυτό. Επίση, πώ βλέπετε το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογία ω καταλήτη για τι μεταρρυθμίσει στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, αυτό, το, αυτό είναι, αφορά αριστεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ερευνών και ε, έρευνα εχμής και χαιρόμαστε πως αυτό το Ερευνητικό Συμβούλιο έχουμε ήδη δύο κατόχους βραβείου Νόμπελ. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να θαρρύνουμε περισσότερη έρευνα, θέλουμε να θαρρύνουμε αριστεία, θέλουμε να έχουμε περισσότερους ε, που έχουν κατόχους βραβείου Νόμπελ. Έγινε ανεξάρτητη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Συμβουλίου, ποιε είναι οι δομέ, ε, οι μηχανισμοί του και η έρευνα ακολουθεί αυτά που αναφέρατε εσείς κύριε Καρβάλιο. Δηλαδή ότι παρόλο που ήταν πολύ επιτυχές έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ιδιαίτερη επιτυχία του Ερευνητικού Συμβουλίου να μπορεί να είναι βιώσιμη στο μέλλον. Υπάρχουν δράσεις που θα πρέπει να αναλυθούν για την δίκησή του, για την τρόπο λειτουργίας του, για τις επιχειρήσεις του και θα πρέπει να ακολουθηθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι κατάλληλες ρυθμιστικές συνθήκες που θα θεσπιστούν για τη λειτουργία του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφορά αριστεία, αφορά αποτελέσματα. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις, όλες τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να στηριχθεί αυτό το Συμβούλιο, για να δώσει αποτελέσματα. Να είστε βέβαιοι ότι η υποστήριξή μου θα είναι αμέριστη όσον αφορά ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαλιάν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Κιγκιάν. Εγώ προερχόμενη από χώρα τη Ανατολική Ευρώπη, θα σα ρωτήσω ακριβώ για την περιοχή μου τι έχετε να πείτε για την έρευνα. Ξέρουμε ότι οι ερευνητέ, οι επιστήμονε στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τα κράτη-μέλη της Κεντρικής και ανατολική Ευρώπη έχουν υψηλότερα εμπόδια θα έλεγα να αντιμετωπίσουν ω προ την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια του 7ου προγράμματο πλαισίου έχουν πιο πολλέ δυσκολίε να, να αναπτύξουν δραστηριότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν, ώστε να αξιοποιήσετε και τα μυαλά ολόκληρη Ευρώπη, που είναι σε όλες τις χώρες Ευρώπη και τη Κεντρική και Ανατολική βεβαίως, έτσι ώστε οι επιστήμονε οι ερευνητέ μα να α, συμμετάσχουν σε έναν ευρύ, διευρυμένο ευρωπαϊκό χώρο έρευνα. Ε, ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστώ, κυρία Βαριάν. για μένα Ευρωπαϊκό χώρος έρευνας είναι και τα 27 κράτη-μέλη. Γιατί είμαι εν γνώση των προβλημάτων που αναφέρατε, είναι πολλά τα προβλήματα και δυσκολίες. Φυσικά είναι πρώτα απ' όλα δύσκολα τα θέματα τα σχετικά με τις υποδομές, όπου μπορούμε να αναλάβουμε δράση αξιοποιώντα τα 26, μέρος των 26 εκατομμύριων ευρώ που προβλέπονται από τα διαφορετικά ταμεία για να αναπτυχθούν οι υποδομέ, αλλά ταυτόχρονα και για να αναπτυχθεί το δυναμικό, οι ικανότητες, γιατί δεν χρειάζονται μόνο υποδομές, αλλά και ανάπτυξη δυνατοτήτων στα μικρότερα κράτη-μέλη, είτε πρόκειται για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, είτε πρόκειται για άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένας ενοποιημένος ευρωπαϊκός χώρος ε, έρευνας θα πρέπει να επιτρέπει τη συνεργασία και των 27 κρατών μελών. Οι υποδομές για την έρευνα, παραδείγματι, το ΕΣΦΡΙ, έχουν ε, επισημάνει, έχουν επιλέξει 44 μεγάλα σχέδια, εκ των οποίων 10 έχουν ήδη αρχίσει την υλοποίησή τους. Ε, καλά παραδείγματα εν μέρη του τι θα μπορούσε να γίνει με μικρές χώρες, Ρουμανία, Τσεχική Δημοκρατία και Ουγγαρία σε μια περίπτωση έχουν ε, συνεργαστεί για την ανάπτυξη υποδομών στον χώρο του λέιζερ, παραδείγματι. Είναι καλά παραδείγματα αυτά. Μικρέ χώρε μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ του. Μικρέ με μεγάλε μπορούν να συνεργαστούν. Και στην αρχική φάση, εκεί που αναπτύσσουμε τι υποδομέ και ε, τι δυνατότητε που, όπω είπα, έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω διακρίσει μεταξύ μεγάλου ή μικρού κράτου μέλου. Όλοι Ευρώπη είμαστε και οι 27 είμαστε Ευρώπη και πρέπει μαζί να συνεργαστούμε στον τομέα της έρευνα αν δεν θέλουμε να εξακολουθήσουμε να χάνουμε τις μεγάλες ευκαιρίες που έχουμε, χάσει, που έχουμε ήδη χάσει και στο παρελθόν. Χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συντονισμό και χρειάζεται να μην φοβόμαστε τη συνεργασία και τον συντονισμό. Η κυρία Βαλιάν έχει συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ. Κύριε Βαλιάν, χαίρομαι που είστε εν γνώση του προβλήματος και πιστεύω και εγώ ότι το θέμα δεν είναι ποιο κράτο είναι μεγάλο ή μικρό, ή αν είναι ένα κράτο μικρό ή μεγάλο για την έρευνά του, γιατί δεν εξαρτάται η έρευνα από τον πληθυσμό. Υπάρχουν χώρε, τι οποίε, όπω είπατε, έχουν προχωρήσει και έχουν θεμελιωθεί ήδη υποδομέ και ικανότητε, ενώ σε άλλε όχι. Χαίρομαι πάντω για την τοποθέτηση σα και ελπίζω ότι θα δούμε στην πράξη ε, εξελίξει και αποτελέσματα κατά την θητεία σας. Ευχαριστώ, κύριος Φαν Ρόι στα αγγλικά. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, μόλι εκφράσατε σαφή άποψη ω προ την ανάγκη να συνεργαστούν τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα πλαίσιο και ενδεχομένω και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πόσο μακροπρόθεσμη μπορεί να είναι αυτή η προσπάθεια, μπορεί να ξεπεράσει τον ορίζοντα του 2013, όπως θα έλεγα εγώ. Ή θεωρείτε ότι πρέπει να ε, είναι μέχρι το 2013. Δεύτερον, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ε, πολύ έδαφος ακόμη να καλύψουν, δεν συμμετέχουν και είναι κρίμα αυτό διότι είναι οι επιχειρήσεις ακριβώς οι οποίες παράγουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα αλλά και θέσεις εργασίας. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν ενδεχομένως στην ενδιάμεση ε, αναθεώρηση του προγράμματος πλαισίου. Και επίσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειαζόμαστε ποσοστώσεις, στόχους, ε, κάποια συγκεκριμένα δηλαδή, κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Διαφορετικά πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια ιδέα από τα όσα έχετε υπόψη σας. Ο τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η ράχοκοκαλιά τη ευρωπαϊκή οικονομία. 25 εκατομμύρια τέτοιε επιχειρήσει έχουμε και είναι το 66% των εργοδοτών στην Ευρώπη. Είναι σημαντική για μα, για όλου μα και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στο πρόγραμμα πλαίσιο. Πώ θα το κάνουμε αυτό θέσατε το στόχο του 15%. Δυστυχώ αυτός ο στόχο δεν επετεύχθη. Είμαστε το 13,4%. Και είναι κρίσιμη προτεραιότητα δική μου να αυξήσω αυτό το ποσοστό από το 13,4% κατά τη διάρκεια της θητείας μου, αν τελικά ε, επικυρωθεί η θέση μου. Μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Μπορούμε να δούμε ε, τι γίνεται όσον αφορά τις, την έρευνα οι έρευνε που γίνονται να ανταποκρίνονται περισσότερο στα ενδιαφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή είναι μια λύση. Και ίσω ε, στα επόμενα προγράμματα εργασία και επόμενες ερεύνες μπορούμε να καθορίσουμε, θα ήθελα εγώ να καθορίσω, στόχο, ε, στόχους, κυρίως με θεματικό τρόπο, δηλαδή εκεί στους τομείς που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να γίνει ευρεία διαβούλευση διότι πρέπει να μάθουμε από τους ε, διάφορους εμπλεκόμενους ενδιαφερομένους τι ακριβώς θέλουν, πού υπάρχουν προβλήματα ε, και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Επίσης πρέπει να τους υποστηρίξουμε όσον αφορά τη δυναμικότητα που δημιουργεί το πρόγραμμα πλαίσιο. Διότι συγχρηματοδοτούμε από κοινού, όπως ξέρετε, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Eurostars που ξεκίνησε πρόσφατα δυνάμει του άρθρου 169 για ε, τεχνολογία εχμής, επιχειρήσεις μικρομεσαίες τεχνολογίας εχμής. Θέλουμε και μέσω του μέσου για τον επιμερισμό του κινδύνου να προσπαθήσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, τους, ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρουν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εχμής, τεχνολογίας εχμής. Ίσως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί πιο ευρέως να συμμετάσχει, αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω. Θέλω μια ομάδα κρούση να δημιουργηθεί, μια task force, αν γίνω επίτροπο, η οποία ομάδα θα εξετάζει αυτό το τομέα. Πού μπορούμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή με το EIF, με τι επενδύσει κεφαλαίων κινδύνου. Uh, μπορούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε περισσότερε μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ο κύριο Βανίστελ Ρόι, ξανά. Κύριε Πρόεδρε, να επανέλθω στο πρώτο τμήμα τη ερώτησή μου. Μπορείτε να πείτε κάτι για τη συνεργασία μεταξύ των ταμείων έχουμε 54 από το πλαίσιο, 86 δις από τα περιφερειακά ταμεία. Λοιπόν, και οι περιφέρειες μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς. Λοιπόν, θέλουμε γνώση, αριστεία που να οδηγεί και στην παραγωγή, ούτω ώστε να ισχυροποιηθεί η Ευρώπη. Μπορείτε να δεσμευτείτε από την πλευρά σας να υπάρξει συνδυασμός ταμείων, πόρων. Το είπατε στην ε, κυρία Βάλια, τη συνάδελφο. Θέλω να δεσμευτείτε για πιο μακροπρόθεσμα πράγματα. Απάντηση. Δεν μπορούμε να πετύχουμε τις πολιτικές που θέλουμε στην Ένωση εάν δεν υπάρξει τέτοια συνεργασία και αν αυτή η συνεργασία δεν είναι συνεχής. Δεν το θεωρώ σαν κάτι καινούριο, ήδη υφίσταται. Το επεξεργαζόμαστε, πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να προωθήσουμε την συνεργασία και αυτό δεν σημαίνει ότι έρχεται το 2013 και ξαφνικά λέμε τέρμα. Αυτό είναι κάτι που και εγώ, αν επιβεβαιωθώ στη θέση μου, αν επικυρωθώ και άλλοι υποψήφοι επίτροποι μαζί μπορούν να εξετάσουν. Υπάρχει τεράστιο τομέα στα διαθετικά ταμεία. Ξέρω καλύτερα τη χώρα μου. Ξέρω πώς χρησιμοποίησαμε τα διαθετικά ταμεία κατά το παρελθόν για να ξεκινήσουμε πολύ φτωχή οικονομία και να φτάσουμε στη τεχνολογία της γνώσης, να φτάσουμε σε μια οικονομία όπου μπορεί να πετυχαίνει πράγματα. Ε, δημιουργήσαμε πλούτο. Αυτό έγινε μέσω σωστή υγιού χρήσεω των διαθροτικών ταμείων, των πόρων των διαθροτικών ταμείων. Και αυτό μπορεί να γίνει και στο μέλλον και σίγουρα θα σα υποσχεθώ ότι εγώ θα υποστηρίξω αυτή την συνέχιση τη συνεργασία συγκεκριμένη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μέρκη, είναι η επόμενη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Με πολύ μεγάλη χαρά ακούω τις δεσμεύσει τι οποίε αναλαμβάνετε για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, γιατί μόνο μία, από δέκα, μία στις δέκα επιχειρήσεις έχει υποστήριξη από το ε, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα αυτή τη στιγμή. Αλλά αφού το καλύψω το θέμα αυτό, περάσω σε κάτι άλλο. Ακούμε, κυρία Γκίγαν Κουίν, πολλά πράγματα για την έρευνα από τα όσα λέτε. Για την καινοτομία όμως, γιατί η καινοτομία δεν εξαντλείται στην έρευνα. Είναι διαφορετική από την έρευνα. Και αυτό το οποίο με ε, ανησυχεί θα ήταν η εμπορευματοποίηση της έρευνας της γνώσης. Η ε, καινοτομία που σημαίνει ταυτόχρονα προσφορά στην αγορά ενός προϊόντος ε, είναι ίσως η δύσκολη πτυχή της έρευνας, γιατί καλοί είμαστε στην έρευνα, καλοί είμαστε στο να, ανακαλύπτουμε νέα, στο να εφευρίσκουμε ενδεχομένω να ανακαλύπτουμε νέα πράγματα, αλλά θα πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να τα διαθέσουμε στην αγορά. Κύριε Κίγκαν Κουίν, βεβαίως σχετίζεται με την αγορά, είναι συνδεδεμένη με την αγορά η καινοτομία και αυτό πρέπει να το ορίσουμε ήδη ο στόχο της έρευνας. Η έρευνα, η εξαίρετη έρευνα που έχει ήδη αναπτυχθεί και που έχει τύχη υποστηρίξεω, πρέπει να φτάσει μέχρι την αγορά, πρέπει να βοηθήσει τι επιχειρήσει που χρειάζονται την έρευνα, πρέπει να επιτρέψει δηλαδή, την πρόσβαση των άλλων στην έρευνα έτσι ώστε και να αντιμετωπίσουμε τι παγκόσμιες προκλήσεις, οικουμενικέ προκλήσει που είναι τα ενεργειακά αισθήματα, η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια επιστηστική, τα προβλήματα στην ε, προσφορά φαρμάκων, ε, η φτώχεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα ε, αντιμετωπίσουμε με τα προϊόντα που θα είμαστε τέλει σε θέση να προσφέρουμε στην αγορά και που θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων και ταυτόχρονα προβαίνοντας αυτή την πορευματοποίηση θα πρέπει να να εξασφαλίσουμε ότι, εξασφαλίσουμε ότι δημιουργούμε μια καλύτερη κοινωνία. Και η καινοτομία, επαναλαμβάνω, δεν είναι ευθύνη ενό μόνο επιτρόπου, ούτε ενό μόνο ημεμονωμένου κράτου μέλου. Είναι μια δραστηριότητα που θα πρέπει σε κάθε επίπεδο οριζόντια να αναπτυχθεί και να στηριχθεί και σε επίπεδο περιβάλλοντος και σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο κρατικό, κοινοτικό, όλοι θα πρέπει να συνεργαστούμε. Να αξιοποιήσουμε την εξαίρετη έρευνα που ήδη υπάρχει και που μπορεί εν τέλει να μας εξασφαλίσει τα προϊόντα που χρειαζόμαστε. Και όπως είπα θα πρέπει να διαλύσουμε τους φραγμούς, είτε πρόκειται για τα πνευματικά δικαιώματα, είτε πρόκειται για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Ε, πρόσβαση στη γνώση, όλοι αυτοί οι φραγμοί πρέπει να αποδιαρθρωθούν για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να παράγουμε καινοτομία. Συμπληρωματικό ερώτημα. Ναι, εσείς ως Επίτροπος Έρευνας και Καινοτομίας, εγώ ανησυχώ, γιατί νομίζω ότι η καινοτομία θα πρέπει να είναι ένα οριζόντιο θέμα στην Κομισιόν. Ευτυχώς έχει πει ο κύριος Παρόσο, ότι η καινοτομία είναι ένα από τους κύριους στόχου τους, από τις μεγαλύτερε προτεραιότητέ του. Και την άνοιξη του 2010 θα παρουσιάσει μια ατζέντα καινοτομία. Πώς σα επηρεάζει αυτό όμως τότε. Θα σας κατευθύνει ο κύριος Μπαρόσο ή θα κατευθύνετε εσείς τους άλλους επιτρόπους. Νομίζω ότι ο κύριος Μπαρόσο θα ήθελε και αυτό να ακούσει την απάντησή μου, λέει η κυρία Γκίγκαν Κουίν. Εάν με επιβεβαιώσετε, αν με επικυρώσετε, θα είμαι ένας ιδιαίτερα δυναμικός επίτροπος. Προφανώς είναι εγκάρσιο θέμα η καινοτομία. Έχω αναφέρει πόσες επιτροπές εμπλέκονται στο θέμα αυτό. Εγώ θα προεδρεύω τη ομάδα των επιτρόπων καινοτομία, ώστε όλοι μα από κοινού να μπορέσουμε να προωθήσουμε την πολιτική καιροτομία για την Κομισιόν και για όλη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μεμονωμένα, αλλά ο καθένας έχει το δικό του τομέα αρμοδιότητα. Είναι ελικρούς που έχει να κάνει με την ψηφιακή, με τα ψηφιακά θέματα, κυρίως και στα θέματα της ενέργειας κτλ. Είναι εγκάσια, σας λέω και πάλι, η αλλά είναι, εξακολουθεί να είναι δική μου αρμοδιότητα να προεδρεύω τη ομάδα καινοτομία στην Κομισιόν και να συνενώνω τι προσπάθειε. Αυτά πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα σφιχτό πλαίσιο. Δεν θέλω επιτροπέ που να μιλάνε και να μιλάνε και να μιλάνε και να μην καταλήγουν σε τίποτα. Θέλω δράση. Θέλω να υπάρξουν στόχοι οι οποίοι θα επιτευχθούν για την Ευρώπη του 2020 και με αυτό το όραμα μπορεί η έρευνα και η καινοτομία να συμβάλλουν στη στατιστική του 2020, του 2020. Θα είμαι λοιπόν συλλογική, αλλά δεν θα είμαι άτομο το οποίο θα κλείνει το στόμα του. Το κύριος Ριβάζη, η κυρία Ριβάζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που ε, θεωρεί τον εαυτό σας σαν μια γυναίκα πολιτικό και ελπίζω να είσαστε ε, μια γυναίκα δράσης που να είσαστε συμβατή με τα οικολογικά Δύο μελανά σημεία βλέπω σημαντικά όσον αφορά τις δημοσιονομικές, ε, τους δημοσιονομικούς προνοτοντισμούς του προγράμματος πλαίσιου. Το πρώτο είναι το πυρηνικό, πυρηνικός τομέας. Αντίθετα με αυτά που υπόθηκαν, ο πυρηνικός τομέας έχει αστρονομικά ποσά τα οποία δίνονται στον πυρηνικό τομέα. 63% του προϋπολογισμού για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας πηγαίνουν εκεί. Και δίνεται μόνο στον πυρηνικό τομέα αυτό το κονδύλι. Και δεύτερον είναι η νανοτεχνολογία θα ήθελα να είσαστε ευαίσθητοι στο εξή. Υπάρχει μια εξέλιξη και διάδοση της νανοτεχνολογίας των νανομόριων και στα τρόφιμα ε, και στα αγαθά τα καταναλωτικά και μόνο 1% του προϋπολογισμού διατίθεται στην αξιολόγηση του κινδύνου. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, είστε έτοιμοι να μειώσετε τα κονδύλια όσον αφορά τον πυρηνικό τομέα και να γίνει ανακατανομή και να αυξηθούν τα κονδύλια πηγαίνουν την αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου για την νανοτεχνολογία. Η κυρία ε, υποψήφια επίτροπο έχει το λόγο. Απάντηση. Δεν θέλω να μειώσω τον προπολογισμό σε κανέναν τομέα ευθύνη μου. Αυτό είναι το πρώτο. Αλλά αυτό θα πρέπει να ειδωθεί. Θα δούμε τι θα γίνει όταν θα συμμετάσχουμε στι συζητήσει, στι λεπτομερεί για τον προπολογισμό. Η πυρηνική ενέργεια για μένα είναι εξαιρετικά σημαντική Um, Απομένει η τεχνολογία ε, της επιλογής πολλών κρατών μελών, δεν παράγει άνθρακα, εκπομπές άνθρακα uh, um, και θα πρέπει να παραμείνει η έρευνα για να αναπτυχθεί ως επιλογή για τα κράτη-μέλη που θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Αυτό που δεν θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να πει στα κράτη-μέλη τι μείγμα ενέργειας είναι κατάλληλο για αυτά αυτό είναι θέμα των κρατών μελών και αυτό αναφέρεται σαφέστατα στη συνθήκη της Λισαβόνα. Και μην ανησυχείτε, εγώ δεν πρόκειται να ανακατευθώ. Ευρατόμ. Ευρατόμ λοιπόν. Πυρηνική έρευνα και δραστηριότητα εκπαίδευση. 2,7 δι στον προπολογισμό και οι τομεί είναι διαχείριση αποβλήτων και ασφάλεια. Αυτό θα συνεχιστεί. Όσον αφορά την νανοτεχνολογία, κάτι που έπρεπε να μάθω, διότι δεν ήξερα πολλά, σχεδόν τίποτα δεν ήξερα για την νανοτεχνολογία, δεν ήξερα καν περί τίνος επρόκειτο. Ενδεχομένε εφαρμογέ τη είναι πάρα πολύ σημαντικέ, όπω είπατε. Είναι σημαντική για τα φάρμακα και για εστιασμένε θεραπείε για τον καρκίνο. Κάτι που αφορά όλου Για την ενέργεια, για αποδοτικέ ηλιακέ κυψέλε, για την χημεία, για καθαρέ χημικές διαδικασίε, διεργασίες. Η νανοτεχνολογία είναι μια τεχνολογία πολύ σημαντική, έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, που σημαίνει περισσότερες θέσεις απασχόλησης για το λαό μας και πολλές από τις θέσεις αυτές αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις. Για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, για μένα δεν είναι θέμα κυρία Ραβάζη να αποφασίσουμε ότι πρέπει να κάνουμε περικοπές από υποστήριξη ενός τομέα για να αυξηθεί υποστήριξη άλλου τομέα. Θα πρέπει να δούμε τον προπολογισμό εν γέννη για τον τομέα και αν είμαι επίτροπος ελπίζω ότι θα μπορέσω να κρατήσω τα κονδύλια όσα έχουν και με την υποστήριξή σας και την υποστήριξη όλων των παρισταμένων να μπορέσουμε να κινηθούμε προς μια διατήρηση των υφισταμένων και ίσως να αυξήσουμε λίγο παραπάνω το ποσά που διατίθενται. Κυρία Ρεβάζη και πάλι. Ναι. Στο πλαίσιο της κρίσης εμπιστοσύνη που έχει ο πολίτης, που νιώθει ο πολίτης στην έρευνα, είστε τετεθειμένοι να στηρίξετε προγράμματα που ε, προτείνει ή ε, περιγράφει η κοινωνία των πολιτών μέσα από το πρόγραμμα ε, πλαίσιο, όπως άλλωστε είχε κάνει και ο προκατοχός σας. Δηλαδή έρευνα που προτείνουν ή καθοδηγούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Απάντηση. Ο κύριος Πορτοτσνίκ, προκατοχός μου, ε, στήριξε και μάλιστα άφησε σημαντικό κληροδότημα, θα έλεγα, σημαντική κληρονομιά. Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχιστεί. Θα στήριχθει, θα αναπτυχθεί περαιτέρω όπου χρειάζεται διότι πιστεύω ότι έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά στον τομέα της έρευνας και δεν θα και εγώ να συνεχιστεί. Θα την υποστηρίξω. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Τουρσνόφσκι έχει το λόγο, ο οποίος κάθεται πίσω σας και θα είναι λίγο δύσκολο να τον δείτε. Είναι αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ κυρία, κυρία Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για την έρευνα, την ε, καινοτομία και εμείς ως μέλη της Επιτροπής Ήτρα, της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στα θέματα αυτά. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο έχετε ήδη θίξει. Θα ήθελα να μιλήσω για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή είναι ο κύκλος καινοτομίας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας, ο κύκλος αυτός είναι κάπως μακρός σε, στην Ευρώπη σε σχέση με τους ανταγωνισμούς μας, ανταγωνιστές μας. Θέλω λοιπόν να διώξουμε αυτή τη γραφειοκρατία η οποία εμποδίζει αυτή την καινοτομία και θέλω τις απόψεις σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, λέει, λέει η κυρία Κίγαν Κουίν. Η έρευνα, η καινοτομία και η επιστήμη έχουν τεθεί από τον Πρόεδρο Μπαρόσο στην καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι ένα ζωτικό στοιχείο για να βοηθήσουμε την Ευρώπη να βγει από την οικονομική κάμψη στην οποία βρίσκεται. Μια πολιτική επίσης η οποία θα προωθήσει την ε, οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανία, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την οικονομική ανάκαμψη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ό,τι πρέπει να γίνει στον τομέα της απλοποίησης και θα επανέλθω στο θέμα αυτό και πάλι και πάλι γιατί είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να κάνουμε <clears throat> και γρήγορα κιόλα για να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε καινοτομία να έχουμε μια σωστή πολιτική καινοτομία που μπορεί να δει η βιομηχανία ότι πράγματι σοβαρά υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια να μεταφέρουμε πόρους στην καινοτομία και στις θέσεις απασχολήσεων, όλα αυτά τα μέτρα της απλοποίησης πρέπει να γίνουν. Είτε είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι <clears throat> για τις κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες, είτε είναι στα κοινά προγράμματα σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα, χρειάζεται να βοηθήσουμε και να εφαρμόσουμε στοιχεία και εργαλεία τα οποία θα προαγάγουν την καινοτομία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Κομισιόν έχει μια ιδιαίτερη σημαντική ευθύνη στον τομέα αυτό να θεσπίσει το ταχύτερο δυνατό τέτοια εργαλεία, να κοιτάξει όλα τα θέματα της καινοτομίας υπό τη δική μου ηγεσία και να θεσπίσει μια εγκάρσια πολιτική που καλύπτει όλους τους τομείς αυτούς, ώστε ό,τι γίνει να γίνει με ένα συνεργατικό και συντονισμένο τρόπο. Ε, έχετε το συμπληρωματικό ερώτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το συμπληρωματικό ερώτημα είναι το εξή. Πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πιο σημαντικά ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη, τον Γαλιλαίο. Πώς μπορεί ο Γαλιλαίος λοιπόν να οδηγήσει σε μια τομή σε ό,τι αφορά την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα. Ο Γαλιλαίος, όπως ξέρετε, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα αλλά είχαμε στο παρελθόν μακρές συζητήσεις, πολλές, ε, πολλούς λογιστικούς ελέγχους, πολλές συζητήσεις για το σύνολο αυτό σχέδιο το Γαλιλαίο. Και τελικά ο κύριος Σταγιάννη, ο οποίος είναι ο αρμόδιος στον τομέα αυτό, είναι αυτός ο οποίος θα συνεργαστεί μαζί μου στην Επιτροπή για την Καινοτομία, στην Επιτροπή των Επιτρόπων για την Καινοτομία, ώστε οι προτάσεις του να ληφθούν υπόψη για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μεγάλο ερευνητικό έργο και την καινοτομία του Γαλιλαίου που χρειάστηκε τόσο χρόνο για να ξεκινήσει, κόστησε τόσο πολύ, που ανησύχησε τόσους πολλοί ιδίω του συναδέλφου του κυρίου Οντή στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί είναι ένα εργαλείο, ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ισχυρό εργαλείο ο Γαλιλαίος, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πολιτική καινοτομία η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της βιομηχανίας, ανταποκρίνεται στα αιτήματα της βιομηχανίας και δείχνει στη βιομηχανία ότι η Ευρωπαϊκή αυτή Επιτροπή θέλει πράγματι να εμπλέξει την βιομηχανία, να κάνει πιο εύκολο να υπάρχει ε, επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη και θέλω να τονίσω ότι εμείς έχουμε προβλήματα αλλά εξακολουθούμε να λειτουργούμε ως επιχειρήσεις και είμαστε έτοιμοι για επενδύσεις από όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας. Η συνάδελφοι τώρα από την Επιτροπή Πολιτισμού ξεκινούμε με τον κύριο Μπόρις. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να σε ευχαριστήσω για όλες τις απαντήσεις που μας δώσατε. Έχουμε μία πρόκληση παγκοσμίων βελίας μπροστά μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ανταγωνιστική οικονομία. Ανταγωνιστική στον κόσμο. Και θέλω να τονίσω τον τομέα της παιδείας. Χρειαζόμαστε να εισαγάγουμε την καινοτομία σαν στοιχείο της παιδείας εν Εξού και το ερώτημά μου, σε ποιο βαθμό προτίθεστε να υποστηρίξετε την παιδεία όσον αφορά αυτό το θέμα, δηλαδή υποστήριξη των οριζοντίων δραστηριοτήτων που αφορούν την πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο, ε, εκμάθηση εξ αποστάσεως, e-learning, ανταλλαγή βελτίστων ε, πρακτικών, υποστήριξη της εκπαίδευσης στον τομέα των επιστημών. Όλα αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν μετά να μεταφραστούν σε ένα καλό επίπεδο παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υποστηρίξετε λοιπόν αυτή την πτυχή της ε, παιδείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι, και ευχαριστώ πολύ κύριε Μπόρις για την ερώτηση σας. Όπως γνωρίζετε, το μέσο της εκπαίδευσης θα ανοίξει το χαρτοφυλάκιο της κυρίας Βασιλείου, της συνυποψηφίου επιτρόπου. Ε, έχουμε συνομιλήσει ήδη, ατύπως, όχι επισήμως, για τρόπους με, τον, με τους οποίους ε, η Επίτροπος ή ο Επίτροπος για την έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει γιατί με την ε, ανακοίνωση της Νέας Επιτροπής ήδη η ήταν υπό την ευθύνη του ε, Πετρόπου για την έρευνα, ο τομέας της έρευνας, τα προγράμματα Marie Curie κτλ. Είναι απαραίτητο λοιπόν πιστεύω να μπει και στην εκπαίδευση ο τομέας της έρευνας ε, τους νέους μας την τελευταία δεκαετία, όπως γνωρίζετε τους έχουμε ενθαρρύνει να αναπτύξουν εμπορικές δραστηριότητες, να αναπτύξουν δραστηριότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Και ξέρουμε τι είδους επιπτώσεις είχαν. Ξέρουμε ότι πια δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό και ότι βρίσκονται υποπίεση θέσεις εργασίας στον τομέα των εμπορικών και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών έτσι λοιπόν πρέπει να πούμε στους νέους μας ότι αν θέλουν να ταξιδεύουν εύκολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουν να αναπτυχθούν στην έρευνα, θα πρέπει κάπως να εστέσουν το ενδιαφέρον, το, τους και γι αυτό, ε, για να έχουν θέσει εργασία. Και γι' αυτό εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να συνδυαστούμε στην ε, επιστήμη και με την κυρία Βασιλείου, εφόσον εγκριθούν οι θέσεις μας, θα δούμε ε, σε ποιους τομείς ο κάθε ένας, το κάθε χαρτοφυλάκιο μπορεί να στηρίξει την πορεία ενός νέου από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια μεταεκπαίδευση τη, μέσα από την έρευνα και όταν θα έχει πια και το πανεπιστημιακό του δίπλωμα τις δυνατότητες που θα προσφέρουμε στο νέο για να βρει θέση εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να μην υπάρχουν τα εμπόδια στην κινητικότητα έτσι ώστε να έχει την ίδια προστασία και για τη σύνταξή του και για την κοινωνική του ασφάλεια, η ασφάλιση και για τις συνθήκες εργασίας του, να ενθαρρύνουμε τους νέους να ασχοληθούν με την επιστήμη και αν μου επιτρέπετε τον άκομψο όρο να καταστήσουμε λίγο πιο σεξι την επιστήμη. Πρέπει να έχουμε πιο πολλούς επιστήμονες. Πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν τους νέους. möchten Sie eine stellen, bitte? Κυρία συνάδελφε, κυρία συνάδελφε, θέλετε να κάνετε μια συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αναφέρεστε επίσης στις προσεχείς χρηματοπιστωτικές ε, προοπτικές. Η επεξεργασία των προτάσεων θα ξεκινήσει το 2011. Ε, υποστηρίζετε την πολιτική συνοχής, η οποία καλύπτει μεγάλο ποσοστό βέβαια των κονδυλίων ε, που πηγαίνουν στην έρευνα. Ποια είναι η θέση σας ως προς την πολιτική συνοχής, ιδιαίτερα για την έρευνα και την ανάπτυξη. Απάντηση. Η συζήτηση για τις ε, επερχόμενες δημοσιονομικές πρόπτικες θα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα και θα έχει μεγάλη δυναμικότητα. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Επιτροπής σας, ακόμα και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του κ. Όντι, για να δούμε τους διάφορους τομείς και να δούμε πώς είναι η καλύτερη κατανομή των κονδυλίων. Και στα πλαίσια αυτά προφανώς είναι πολύ σημαντική η πολιτική συνοχή. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποια χώρα να υπολείπεται <clears throat> των υπολείπων. Όλοι πρέπει από κοινού να προχωρήσουμε και για να το κάνουμε αυτό είναι πάρα πολύ ζωτικός ο ρόλος της συνοχής. Και εγώ πιστεύω ότι η έρευνα πρέπει να εμπλέκεται κεντρικά σε οποιαδήποτε μορφή πολιτικής συνοχής. Να είσαστε σίγουροι ότι εγώ θα εργαστώ με τους συναδέλφους μου, εάν με ε, επιβεβαιώσετε για να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι κάνουμε θα γίνει με ένα συνεργατικό και συντονισμένο τρόπο ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε. Το τι θα γίνει τώρα στις δημοσιονομικές προοπτικές, αυτό βέβαια είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπάντια Ικουτσέ έχει το λόγο. Ελπίζω ότι το προφέρω σωστά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι είπατε ότι έχετε ίδια σε επαφή με την κυρία Βασιλείου, η οποία είναι υποψήφια επίτροπος παιδείας και κουλτούρας, διότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια κοινή δράση και στον τομέα της έρευνας και της κατάρτισης. Η έρευνα είναι ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης και ευμάρειας, είπατε, ότι θέλετε να θεσπίσετε μια σαφή στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης με στόχο η στρατηγική 2020 να μπορέσει να καρποφορήσει. Εγώ θα ήθελα να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι συγκεκριμένες δράσεις ή δυνατόν και πώς θα ε, εξασφαλίσετε την αναβάθμιση των προσόντων των εργαζομένων αν χρειάζεται να προωθήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία έχουν σαν στόχο την καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων έναντι των αναγκαιότητων που προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ευχαριστώ, <clears throat> κυρία Γίγαν Κουίν. Νομίζω ότι καταρχάς θα έπρεπε να συμφωνήσω με το σχόλιο που κάνατε, ότι είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη έρευνα και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το 2020 η έρευνα διαδραματεί σημαντικότατο θεμελιώδη ρόλο. Αλλά το πρόγραμμα αυτό θα είναι υπό την ευθύνη της κυρίας Βασιλείου αυτό που αναφέρατε. Όμως θα εφαρμοστεί από τον εκτελεστικό φορέα για την έρευνα που θα τελεί υπό τη δική μου ευθύνη και αυτό βεβαίως είναι θέμα που καλύπτει τη δίκηση και την εκτέλεση των, διαχείριση και εκτέλεση των προγραμμάτων. Εκείνη θα είναι υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, τις κοινότητες για τεχνολογία και τη γνώση και είναι αν θέλετε τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με συντονισμένο τρόπο, ούτω ώστε να πετύχουμε τα αποτελέσματα αυτά που αναφέρατε. Οι ερευνητικές πολιτικές όσον αφορά τα πανεπιστήμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα πόσο στο τμήμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που θα παραμείνει δικός μου τομέας ευθύνη. Άρα είναι πολύ σημαντικό και ένα από τους λόγους για τις άτυπες συζητήσεις που ήδη έγιναν είναι πολύ σημαντικό λέγω ότι και να κάνουμε ό,τι κάνει εκείνη και εγώ να είναι συμπληρωματικά, να συμπληρώνονται οι δύο πολιτικές. Δύο πολιτικές που λειτουργούσαν από κοινού μέχρι τώρα, που κατά κάποιο τρόπο έχουν διαχωριστεί, να εξακολουθήσει η συνεργασία όταν, όπως όταν ανήκαν σε μια γενική διεύθυνση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν έχουμε καλή σχέση επικοινωνίας μεταξύ μας. Έχουμε 4.000 ε, τριτοβάθμια ε, φορείς με, ε, με 7 εκατομμύρια ε, φοιτητές. Δεν συμμετέχουν αρκετοί από αυτούς τους φορείς έρευνα Μπορούμε λοιπόν και οι δύο μαζί να συνεργαστούμε, να ενθαρρύνουμε περισσότερους φορείς τριτοβάθμιους να ασχοληθούν με την έρευνα. Διότι μόνο 33 από τα πανεπιστημιακά δήματα της Ευρώπης είναι στο 100 πρώτα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Όπως είπατε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάρα πολλοί παίκτες μέσα σε εισαγωγικά οι οποίοι εμπλέκονται στο θέμα αυτό. Εγώ θα ήθελα να γνωρίσω πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να επιτύχετε μια συμφωνία, μια συνένεση μεταξύ όλων αυτών των εμπλεκομένων ώστε να καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια ώστε πραγματικά η κατάρτιση των εργαζομένων, των νέων φοιτητών να είναι επιτυχής για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να τους ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν σε αυτόν τον τομέα της παιδείας. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν έχουν μπει όλοι σε αυτόν τον τομέα της εκπαίδευσης, δεν συμμετέχουν αρκετά, πρέπει να τους αποδείξουμε ότι είναι ένας τομέας όπου στο τέλος της εκπαίδευσής τους μπορεί να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, να βρουν μια δουλειά, να απασχοληθούν να χρησιμοποιήσουν την εκπαίδευσή τους και την κατάρτισή τους για να πάνε και στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να εργαστούν όπου επιθυμούν. Αυτό είναι σημαντικό να ρυθμιστούν όλα αυτά που προανέφερα. Το θέμα συνταξιδοτικών δικαιωμάτων, συνθήκες εργασίας και διαμονής. Πρέπει να τα κάνουμε αυτά σε στενή συνεργασία μεταξύ μας. Δεν ξέρω επιμακρών την κυρία Βασιλείου, αλλά νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να συνεργαστώ στενά και δεν έχουμε επιλογή νομίζω αυτά τα θέματα σε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν γέννη. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ διαφόρων επιτρόπων. Δεν μπορούμε πλέον να, να εργαζόμαστε απομονωμένα. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, ιδιωτικές επικράτειες. Ε, Βασίλεια. Πρέπει να εργαζόμαστε αποτελεσματικά συντονισμένα μαζί, ούτω ώστε να δώσουμε αποτελέσματα. Πολιτική που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα που περνάμε οικονομική κρίση που περνάει η κρίση οικονομική όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το κάνουμε αυτό, μπορεί να αποτελέσματα για την Ένωση. Και από τη δική μου πλευρά, εγώ προτίθεμαι να εξασφαλίσω ότι θα πετύχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο παπα Παπα-Νικολάου από την Επιτροπή Πολιτισμού επίση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν και προηγουμένω. Πολλοί είναι εκείνοι οι νέοι επιστήμονες οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους με έρευνα και γι' αυτό αποτελεί καθήκον όλων μας να διασφαλίζουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για εκείνους έτσι ώστε να αποτρέψουμε και τη διαρροή εγκεφάλων από τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνα, που αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δεδομένο που πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μα, και βεβαίω να καταφέρουμε να προσελκύσουμε λαμπρού επιστήμονε που βρίσκονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι ε, εκ των πραγμάτων έχουν μόνο θετικά να συνεισφέρουν στην προσπάθεια την ερευνητική της Ευρω... σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς σκοπεύετε να προωθήσετε τα παραπάνω ζητήματα, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή έρευνα στερείται ικανών πόρων χρηματοδότησης και το λέω αυτό αναφέροντας συγκριτικά τους στόχους της Λισαβόνας. Ε, όλοι θυμόμαστε ότι 3% του ΑΕΠ ήταν το, ο επιδιωκόμενος στόχος. Τελικά το ε, επίπεδο που καταφέραμε να φτάσουμε ήταν μόνο το 1,9%. Πώς νομίζετε ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών στη χρηματοδότηση θα μειωθούν και πώς θα καταφέρουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των νέων ερευνητών, ε, των λαμπρών αυτών επιστημόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Εάν θέλουμε, λέει η κυρία Γίγαν Κουίν, αν θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους επιστήμονες και τους ερευνητές στην Ευρώπη, και έχω απόλυτη επίγνωση της διαρροής των εγκεφάλων, θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες εργασίες που κάνουν ελκυστική την Ευρώπη και ελκυστική την παραμονή των ερευνητών εδώ. Αυτές, αυτές οι συνθήκες εργασία μπορεί να άπτονται των θεμάτων που ανέφερα προηγουμένως για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα τι συνθήκε εργασία, αλλά επίση, και να άρουμε του φραγμούς στα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων, το τομέα των ευρεσιτεχνιών, δηλαδή των προβλημάτων που κάνουν πολύ πιο δύσκολη τη μεταλαμβάνευση τη γνώση από του ερευνητέ αυτού. για το στόχο του 3%. Το 3% είναι ένα θέμα θλιβερό, αν θέλετε, ότι το γεγονό ότι δεν φτάσαμε ακόμα αυτό το στόχο του 3% και είδαμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ομπάμα, είπε ότι και αυτό έχει αυτό το στόχο Πρέπει να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε στα θέματα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε σε τελμάτωση ακόμα στο 1,85%. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι η αιτία αυτού του φαινομένου. Πού θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας και πώς. Αν δούμε λοιπόν ότι <clears throat> υπάρχουν και δύο συνιστώσεις, η δημόσια και η ιδιωτική συνιστόσα της χρηματοδότησης, είναι απαραίτητο ότι πρέπει να προωθήσουμε και μια αύξηση στην ιδιωτικά χρηματοδούμενη έρευνα μόνο με την άρση των φραγμών, των οδοφραγμάτων, των δυσκολιών, με την απλοποίηση, με όλα τα μέσα στη διάθεσή μας, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι μεγάλες επιχειρήσεις, είτε είναι πολυεθνικές εταιρείες. Θα πρέπει να άρουμε λοιπόν όλους τους φραγμούς και τα σημεία συμφόρησης, τα οποία εμποδίσουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα και αυτό είναι μια τεράστια προτεραιότητα για μένα. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το στόχο του 3% Ορισμένοι λέγανε σε δημοσιεύματα στον τύπο ότι πρέπει να μειώσουμε αυτό. Αυτό θα ήταν το λαθασμένο μήνυμα. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να αυξηθούν οι δαπάνες αυτές και είναι δύσκολο σε χρόνο οικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ πολύ Λεωπρόεδρος, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα βλέπω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να ξεπερνάμε το χρόνο μας. Ενώ είχαμε ξεκινήσει πολύ καλά ως προς το χρόνο, τώρα σιγά σιγά δυσκολεύει η κατάσταση. Και παρακαλώ τον κύριο Γιόρνταν Σίζελ να λάβει το λόγο. Την κυρία Γιόρνταν Σίζελ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Για να επανέλθω στην καινοτομία. που στο επίκεντρο και τη φυσταμένη στρατηγική Λισαβόνα, αλλά και τη νέα ασφαλώ 2020, 2020 Πολλές φορές μιλάμε για την έρευνα, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και την καινοτομία ως προς τους όρους, τους κοινωνιολογικούς, τα θέματα τα οργανωτικά. Και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις ως προς μια ολιστική προσέγγιση στην καινοτομία. Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε καλές ιδέες και να τις προστατεύσουμε ταυτόχρονα, γιατί πρέπει να υπάρξει και οικονομική υποστήριξη αλλά και οι ανθρώπινοι πόροι για να εξασφαλιστεί, για να αναπτυχθεί η καινοτομία. Οποιαδήποτε λοιπόν σχετικά μέτρα, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, ε, θα πρέπει να βλέπει και τη σχετική ανταμοιβή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε σήμερα ότι τα αποτελέσματα τα οποία αναμένονται στο τομέα αυτών δεν θα, είναι, δεν θα τεθούν σε κίνδυνο ε, από κάποιες άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απάντηση. Η πολιτική για την καινοτομία είναι κατ' ουσίαν η διασφάλιση του ότι οι νέες εφευρέσεις, οι νέες ανακαλύψεις, ε, η νέα γνώση που παράγεται μπορεί να διατεθεί στην αγορά και να ικανοποιήσει ανάγκες που έχει η Ένωση και τα προϊόντα αυτά που διατεθεί στην αγορά ταυτόχρονα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, τις συνθήκες διαβίωσης ε, γιατί βεβαίως με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής χρειαζόμαστε ε, καλύτερα προϊόντα στον τομέα αυτών, είτε τη στήριξη ε, ε, του ανθρώπου στην διαβίωσή του, είτε καλύτερα φάρμακα, είτε σχετικό εξοπλισμό. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα καταφέρουμε και εμείς οι πολιτικοί και οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές προσδιορίζοντα κοινού στόχου, ένα θα είναι ο κύριο κοινό στόχο, ότι δηλαδή ε, θα προσδιορίσουμε, το πώς θα προσδιορίσουμε την καινοτομία ίσως οι πολιτικοί να έχουν μια δική τους έποψη και οι υπόλοιποι, όλοι οι υπόλοιποι να βλέπουν τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Αλλά πάλι υπάρχει κοινό πεδίο νομίζω, πάνω στο οποίο θα πρέπει να στηριχθούμε και να θεμελιώσουμε την ε, έρευνα και την κοινοτομία. Δηλαδή έρευνα, επένδυση καλύτερα στις ε, οικολογικές επενδύσεις, στην οικολογική καινοτομία, τεράστιες προκλήσεις για την Ένωση αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, στις οποίες θα πρέπει να διαθέσουμε τους απαραίτητους πόρους, να επενδύσουμε, να εξασφαλίσουμε την παρουσία και συμμετοχή και των μικρομεσαίων αλλά και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτών. Ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημασία που έχουν, τη μεγάλη σημασία που έχουν οι νέες ιδέες και να προσφέρουμε και την απαραίτητη στήριξη ανθρώπινοι και άλλοι στην αξία αυτή που είναι οι νέες ιδέες. Και να έχει ο ερευνητή που παράγει νέα γνώση, τη στήριξη που θα είχε και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα δραστηριοποίηση επαγγελματική, επιχειρηματική ή άλλη. Ah, um, um, Κοιτάξτε, έχω να κάνω μια δεύτερη ερώτηση όσον αφορά ε, αυτό που ετοιμάζει η Γενική Διεύθυνση Επιχείρηση για την Καινοτομία και ελπίζω να πετύχετε να συντονιστεί η Γενική Διεύθυνση Έρευνα και η Γενική Διεύθυνση για τι Επιχειρήσει. Αυτή η πρόταση θα πρέπει να δημοσιευτεί πριν την άνοιξη φέτο. Θα προτείνετε να έρθει πιο κοντά αυτή η προθεσμία ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατόν να πετύχουμε ε, το στόχο του 2020 και τη στρατηγική για την καινοτομία. Η στρατηγική του 2020 είναι για να ανοίξει ένα δρόμο για να βγούμε από την κρίση και να δημιουργηθεί μια ε, οικονομία βιώσιμη, ε, οικονομία κοινωνικής μορφής. Η, αυτή η πρόταση για την καινοτομία, όπως είπατε σωστά κύριε Σιζέλη, είναι ένα σημαντικό στοιχείο ε, του προγράμματο εργασία τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω, αυτό το πρόγραμμα εργασία δεν υιοθετήθηκε ακόμα και είναι πολύ νωρί να συζητήσουμε τον χρονισμό τη πρωτοβουλία. Δεν αμφισβητώ την υλοποίηση τη πρωτοβουλία. Το μόνο που αμφισβητώ σε αυτή τη φάση είναι κατά πόσο πρέπει να γίνει αυτό τότε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να υποβληθεί μια πρόταση στην καινοτομία, να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι ενδιαφερόμενοι. Έγινε αυτή η διαβούλευση για εκεί της, της 2020 που ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Έγινε και συζήτηση δημόσια για την πολιτική καινοτομία. Ε, τώρα θα πρέπει να υποβληθεί η πρόταση. Είναι στο πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι πολύ πρόημο τώρα να σα πω ακριβώ πότε θα γίνει, πότε θα υποβληθεί αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Κορέα Ικάμπου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρία Γκιόγεν Κουίν, ο πρόεδρος Μπαρόσο ενώπιον του κοινοβουλίου μας, δήλωσε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια επανάσταση στην έρευνα και την καινοτομία για μια κοινωνία πληροφορίας. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει τεράστιο γραφειοκρατικό άχθος. Η δυσαρέσκεια του επιστημονικού κόσμου και η διστακτικότητα της βιομηχανίας για τα οποία υπάρχουν πολλοί σαφής, σα, σαφή στοιχεία, μας δείχνουν ότι υπάρχει μείωση του ενδιαφέροντος των εμπλεκομένων. Πώς θα ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Θα είναι επαρκής μία βελτίωση εργαλείων που στο παρελθόν δείχτηκαν να είναι αναποτελεσματικά για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020. Μήπως πρέπει να έχουμε <clears throat> στόχους πολιτικούς και χρηματοοικονομικούς Πώς θα πείσουμε τα κράτη-μέλη να επιτύχουν το στόχο του 3% για την έρευνα και την ανάπτυξη και πώς θα, συμβιβαστεί, πώς θα συναρμοστεί αυτή η πολιτική με την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ η κυρία Επίτροπος. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για κάποιον που είναι απλώς υποψήφιος επίτροπος να αρχίσει να μιλάει για benchmarks και χρηματοδότηση και επίτευξη των στόχων σε λεπτομεριακό επίπεδο. Μπορώ να σας πω όμως το εξής. Όλα αυτά είναι ένα κομβικό και σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής 2020 και βρίσκονται στην καρδιά της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετέθηκαν εκεί από τον κύριο Μπαρόζου. Είναι ρόλος μου και καθήκον μου να πραγματοποιήσω αυτή την πολιτική μέσα στην Κομισιόν. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με συνεργασία, με καλύτερο συντονισμό, με κοινή δράση για να επιτύχουμε <clears throat> την υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Υπάρχουν τομείς στην απλοποίηση των υφισταμένων δομών που θα πρέπει να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό. Έχουμε κάνει πολλά, είναι πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν. Το να με βοηθήσετε να καταλάβω τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αυτό είναι απόκειται στη δική σας επιτροπή και στην ε, ενδιάμεση αξιολόγηση που θα γίνει του προγράμματος πλαισίου 7, εγώ <clears throat> δεν γνωρίζω ποια είναι αυτή η αξιολόγηση. Τώρα ξεκινάει το έργο της η Επιτροπή Αξιολόγηση τον επόμενο μήνα, αλλά εγώ θα ατενίσω πολύ προσεκτικά τις προτάσεις και θα αξιολογήσω τις προτάσεις που περιλαμβάνουν σε αυτή την ενδιάμεση αξιολόγηση. Γιατί πιστεύω ότι θα μας δώσει ένα οδικό χάρτη, θα καταλάβουμε πού είναι τα σημεία συμφόρησης, πού είναι τα προβλήματα όπου πρέπει να επέλθουν αλλαγέ, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πολιτική καινοτομία που να περιλαμβάνει όλους τους επιτρόπους που είναι αρμόδιοι, είτε είναι βιομηχανική καινοτομία, είτε είναι ψηφιακή καινοτομία, είτε είναι καινοτομία στο επιχειρήν. Θα πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι πτυχές σε μια εγκάσια ε, συνεργασία να καταλήξουν σε μια κοινή πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συμπληρωματικό ερώτημα. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, στην απάντησή σας στο γραπτό ερωτηματολόγιο είπατε ότι θα χρησιμοποιήσετε το κοινό κέντρο ερευνών για τον καθορισμό πολιτικών που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών χαμηλής χρήσης άνθρακος γνωρίζοντας ότι υπάρχουν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, θεωρείτε ότι τα κοινά κέντρα ερευνών είναι τα καλύτερα, τα πιο πρόσφορα εργαλεία για να γίνει αυτή η κίνηση προς νέες τεχνολογίες χαμηλού άνθρακος. Νομίζω τα κοινά κέντρα ερευνών είναι σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα <clears throat> για να έχουμε έρευνα που είναι ανεξάρτητη, που είναι σεβαστή από τους άλλους και η οποία χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία και από τα κράτη-μέλη, επειδή <clears throat> οι τελευταίοι είναι πεπισμένοι για την ανεξαρτησία αυτής της έρευνας, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα κοινά κέντρα ερευνών δεν ανήκουν σε κάποιο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ή βιομηχανικό φορέα. Δεν διαφεντεύονται από ομάδες πίεσης. Είναι πηγές ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνη που έχουν χρησιμοποιηθεί και από τη βιομηχανία και από την ίδια την Κομισιόν. Η έρευνά τους είναι πολύ χρήσιμη για τη χάραξη πολιτικής σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει αυτή η πορεία και έχετε την πλήρη μου δέσμευση ότι εγώ θα συνεχίσω να υποστηρίζω την ανεξαρτησία των κοινών και Ευχαριστώ. Ο κύριος Σον Κέλλη έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα όσα επιτύχατε στην πολιτική σαδηροδρομία από την ε, μέρα που διαδεχθήκατε τον πατέρα σας μέχρι σήμερα. Είπατε και παραθέτω, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει τομέα αριστεία στην έρευνα, την κοινοτομία και την, επιστήμη. Και, την επιστήμη. και χαίρομαι που είπατε το, τις λέξεις μπορεί να γίνει. Γιατί από τον ΩΣΑ η περσινή έκθεση δείχνει μια μάλλον ε, φαιά εικόνα, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση επί του ΑΕΠ της ε, δαπανά μόνο 1,77% για την έρευνα. 2,6 Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία το διπλάσιο 3,54%. Έτσι λοιπόν, ε, και ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλήσει μεταξύ των κρατών μελών τη ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Σουηδία, η οποία έχει το 3,6% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ τη, η Ιρλανδία έχει 1,3% μόνο και ορισμένες χώρες μόνο κάτω από το 1% του ΑΕΠ του δαπανούν για την έρευνα και τεχνολογία. Για να δημιουργηθούν λοιπόν τέτοιε θέσει εργασία όπω αυτέ που προβλέπετε, με αυτέ τι ωραίε λέξει, τεχνολογία και οικονομία τη τεχνολογία, η ευφυά τεχνολογία, θα ήθελα να μα εξηγήσετε πώ θα μπορέσουμε να καλύψουμε το χάσμα που ε, μα χωρίζει από τι ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Απάντηση. Καταρχάς νομίζω θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ως, σημαντικότερο, ως τον σημαντικότερο εταίρο της Ευρώπης για την έρευνα και τεχνολογία της Ηνωμένες Πολιτείες και για, την αμοιβαία, ε, για τις αμοιβαίες επενδύσεις και για τις ροές επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ των δύο κρατών ή ενωτήτων ε, και για τον όγκο των κοινών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουμε και για τον, ε, για τον όγκο, τον αριθμό των κοινών μας δημοσιεύσεων. Είναι ο κύριο λοιπόν εταίρο μα στο πρόγραμμα πλαίσιο. Στρατηγικέ εταιρικέ σχέσει έχουμε και με τις ΗΠΑ όντω σε διάφορου τομεί, όπως Task Force, ε, ομάδα κρούσης Ευρωπαϊκής Ένωσης των ΗΠΑ ε, για την βιοτεχνολογία, η Ενεργειακό Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης των ΗΠΑ που θεσπίστηκε πριν από μερικούς μήνες. Ωστόσο, θα πρέπει το όντι να ενισχύσουμε αυτές τις δραστηριότητες περαιτέρω, τις υφιστάμενες δομές, ε, όπου υπάρχουν, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες δομές προς όφελός μας και δομές που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της συνεργασίας. Και αν κοιτάξουμε τα ψυχρά στοιχεία ε, και συγκρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία φετέρου αλλά και άλλους μεγάλους ε, παράγοντες όπως Ινδία, Βραζιλία κτλ. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση να φαίνεται σχετικά σε δυσμενή θέση έναντι των μεγάλων αυτών εταίρων και παραγόντων σε όλο τον κόσμο και θα πρέπει να συναγωνιστούμε μαζί τους αλλά και να συνεργαστούμε μαζί τους μέσα από τις υφιστάμενες δομές είτε με ανάπτυξη νέων δομών, όπως πρόσφατα έγινε με τη θέσπιση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για την ενέργεια. Και αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να, σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να αναλυθούμε. Για δε τους στόχους ε, τους προσωστιαίους επί του ΑΕΠ, το στόχο του ΑΕΠ, του 3%. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρω τον τρόπο να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη και τον ιδιωτικό τομέα να αναζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα ε, αυξηθούν οι δαπάνες. Φυσικά, ε, όταν ε, επικρατεί οικονομική κρίση, η αντίδραση αυτόματη ίσως να είναι να μειωθούν οι δαπάνες για την έρευνα και τεχνολογία. Πράγμα όμως το οποίο ε, δεν έκανε η Φινλανδία πριν από μερικά χρόνια και το αποτέλεσμα είναι ότι τώρα βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Είναι σε επίπεδα αντίστοιχα με τη Σουηδία αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και τους άλλους να το πράξουν αυτό. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Μας είπατε ότι ελπίζετε να εξασφαλίσουμε ένα πρόγραμμα έρευνας που θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Πιστεύετε ότι πράγματι σε πέντε χρόνια θα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτή σας την πρόβλεψη ή θα αποδειχθεί μια ουτοπική μόνο επιθυμία. Απάντηση. Το πρόγραμμα πλαίσιο, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο με δημόσια χρηματοδότηση ερευνητικό πρόγραμμα του κόσμου και ελπίζω, διατηρώ την ελπίδα ότι από τώρα και μέχρι το τέλος της θητείας μου, εφόσον ε, επικυρωθεί η επιλογή μου, η εκλογή μου, ε, δεν θα συμβεί τίποτε το οποίο να ανατρέψει την πρόβλεψη αυτή. Ότι το προσεχές δηλαδή πρόγραμμα πλαίσιο θα είναι σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα και θα ε, αποδειχθεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ε, έρευνας με δημόσια χρηματοδότηση. Γιατί αν κοιτάξουμε τα ποσοστά, αν δούμε τα ποσά της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατικά, Έχουμε να κάνουμε 246 δισεκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και τεχνολογία στην Ευρώπη. Τεράστια θα Ξέρω ότι ο κάθε ερευνητής και ο κάθε επιστήμονας θα σα πει Μα δεν φτάνουν. Ναι, βεβαίω και δίκιο θα έχει. Σωστά θα το πει. Αλλά το πρόγραμμα πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή με την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση που θα γίνει στου επόμενου δύο-τρει μήνες ε, θα μου επιτρέψει εμένα να το κοιτάξω πολύ προσεκτικά, κύριε Κέλλη, ω προ το πώ διδασκόμενοι από τα όσα θα διατυπωθούν ως παρατηρήσεις για το, Ευρωπαϊκό, για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ε, αλλά ταυτόχρονα και αν επικυρωθεί η εκλογή μου, πιστεύω ότι και εγώ και η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας θα έχουμε χάρη σε αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση την ευκαιρία να θεσπίσουμε τις αλλαγές που θα χρειαστούν για το προσεχές πρόγραμμα πλαίσιο, τις αλλαγές που θα χρειαστούν, τις μετατροπές, τους, ε, τις δομές, την απλούστευση που θα χρειαστεί. Κύριος Ράνστορφ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ιστορικά η φτηνή εργατική δύναμη ήταν εμπόδιο στην καινοτομία. Έχουμε τέτοια παραδείγματα πολλά από το παρελθόν. Τώρα που βρισκόμαστε σε μια βαθιά κρίση, αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο και η ευρωπαϊκή παραγωγή να μετεγκατασταθεί σε χώρες με, φτηνά, με φτηνό εργατικό δυναμικό όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, η Αφρική, η Λατινική Αμερική. Πώς σχεδιάζετε λοιπόν να αντιμετωπίσετε αυτό το κίνδυνο ή να μειώσετε εν πάση περιπτώσει αυτό το κίνδυνο. Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το κίνδυνο με την εγκατάσταση της βιομηχανικής μας δραστηριότητα σε χώρες με φτηνότερα εργατικά χέρια. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα αυτό, λέει η κυρία Γκίγαν Κουίν. Γιατί δεν εμπλέκει μονάχα εμένα, αν επικυρωθεί ο διορισμό μου, αλλά και πολλού άλλου στην Κομισιόν και άλλου τομεί πολιτική όπου πρέπει να εργαστούμε από κοινού. Αυτό που κάνουμε σήμερα στον τομέα τη έρευνα, έχουμε αναγνωρίσει το ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί ανταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο που δεν περιμέναμε πολλές φορές να είναι ανταγωνιστές μας σήμερα, όπως η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία, η Ιαπωνία. Και υπάρχουν πολλοί τομείς που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να δούμε τι κάνουμε στους τομείς αυτούς. Συνεργαζόμαστε με τη Βραζιλία στον τομέα των βιοκαυσίμων. Συνεργαζόμαστε με την Ινδία για την ηλιακή ενέργεια, με την Κίνα σε ό,τι αφορά την αεροναυπηγική. Πρέπει να είμαστε αρκετά ανοιχτοί για να κατανοήσουμε ότι αυτοί είναι πραγματικοί ανταγωνιστές που δεν μπορεί, να μπορεί πριν από 10-12 χρόνια να μην ξέραμε ότι θα είναι εδώ μπροστά μας, αλλά σήμερα είναι ενώπιόν μας, είναι πολύ αποτελεσματική, πολύ κινητική, πολύ επιθετική. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, ώστε σε τελική ανάλυση να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπολοιπόμεθα αυτών των ανταγωνιστών στο μέλλον. Υπάρχουν τομείς όπου έχουμε υστερήσει εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών όπως η Ινδία, τα θέματα της ενοτεχνολογίας. Παραδείγματο χάρη, είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε μια συνεργασία και να επενδύσουμε στους τομείς που είναι απαραίτητο για να μην βρεθούμε πίσω από τους ανταγωνιστές μας. Συμπληρωματικό ερώτημα. Σας ευχαριστώ. Η πρόσφατη κρίση είναι ένα ακόμα ε, μια απόδειξη της θεωρίας των μεγάλων κύκλων του Κοντράτιεφ. Τι έχετε κάνει για να δημιουργήσετε συμπλέγματα καινοτομία σε μια τέτοια κατάσταση που είναι τόσο πολύπλοκη. Αν δούμε το άρθρο 169, έχουμε ήδη δημιουργήσει συμπλέγματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το σχέδιο Bonus, το οποίο αφορά τη Βαλτική και μία σειρά από χώρες που βρίσκονται στην περιφέρεια της Βαλτικής θάλασσας, που συνεργάζονται για όλα αυτά τα θέματα τα οποία εμπλέκονται στον χώρο της Βαλτικής. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ένας άλλος χώρος είναι αυτός τον οποίο ανέφερα προηγουμένως, α, <clears throat> νομίζω στην κυρία Βάλεα, είπα ότι όταν έχετε μικρότερες χώρες οι οποίες συνεργάζονται σε ένα σύμπλεγμα, σε ένα κλάστερ, σε έρευνα για θέματα που καμία από αυτή θα μπορούσε από μόνη της μεμονωμένα να καλύψει, είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε λοιπόν όλους αυτούς τους ερευνητικούς χώρους και με τον τρόπο αυτό θα έχουμε εργαλεία που θα είναι χρήσιμα σε όλους μας, είτε θα είναι στο πλαίσιο του προγράμματος πλαίσιο 7, είτε για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ερευνητικού χώρου, είτε στον τομέα της απλοποίησης και της εξασφάλισης ότι η Ευρώπη είναι ένας ζωντανός οικονομικός χώρος. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαραίτητο να γίνουν με πολιτικές οι οποίες θα καρποφορήσουν τελικά. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο ο κύριος Ρόντε, ο οποίος βρίσκεται στα πίσω, βρίσκεται πίσω σας, από την άλλη πλευρά όμως. Καλώς ήλθατε στην Επιτροπή μας. Είναι πάντα χρήσιμο να έχουμε μια υποψήφια επίτροπο η οποία έχει σαφείς απόψεις και σαφήνες σε αυτά που λέει. Μπορείτε να μου δώσετε και εδώ ίσως μια σαφή απάντηση. Έχετε κάποιες εγγυήσει από τον κύριο Μπαρόσο ότι θα χρήξει πράγματι νέα χρήματα στον χώρο της έρευνας τα επερχόμενα χρόνια. Θα με σκοτώσετε με αυτά που λέτε. Κύριε Ρόντε, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Μπαρόσο εφόσον δεν θα έχει μια νέα επιτροπή παρά μόνο μέχρι το τέλος των ακροάσεων, ξέρετε δεν μπορεί να δώσει καμία εγγύηση σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Όλα αυτά θα αρχίσουν να γίνονται σαφή όταν μπούμε στη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές, όταν ξεκινήσει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και σας είπατε θα είναι εύκολες αυτές οι συζητήσεις <clears throat> από πολλές απόψεις και για τον δικό μου τομέα αρμοδιότητας, αν εγκριθώ από το Κοινοβούλιο, θα χρειαστώ την ισχυρή σας υποστήριξη για να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε και ενδεχομένως να το αυξήσουμε. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει και μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των μελών της Κομισιόν για να αποκτήσουν την υποστήριξη που θέλουν ο καθένας για τον τομέα του. Επομένως, ο κύριος Μπαρόσο δεν έχει κάνει καμία δέσμευση σε σχέση με τα χρήματα τα οποία θα δοθούν ε, στο μέλλον στον τομέα αυτό. Και όπως ξέρουμε, λέει ο κύριος Ρόντε, τα χρήματα δεν ακολουθούν την καλή θέληση, γι' αυτό πρέπει να επανέλθω στο, στην απάντησή σας στην κυρία Ριβάση. Είπατε ότι δεν θέλετε να περικόψετε κανένα τομέα αρμοδιότητό σας. Αυτό σημαίνει δεν θα έχετε νέα κατανομή προτεραιοτήτων μέσα στο χαρτοφυλακείο σας ότι δεν θα διαπραγματευτείτε καμία μετακίνηση χρημάτων από μία περιοχή σε μια άλλη. Αν έτσι έπρεπε δεν χρειάζεται να έρθουμε σε αυτή την ακρόαση. Λυπάμαι αν έδωσα τέτοια εντύπωση απαντώντα στην ε, κυρία Ριβάση. Πάντω, σε κάθε τομέα δραστηριοτήτων, σε κάθε δημοσιονομικό τομέα πρέπει να καταγράφεται τι φέρνει αποτέλεσμα, καλό, τι φέρει ένα μέτριο αποτέλεσμα και τι χρειάζεται να ε, αλλάξει άρδιν. Πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει μόνο όταν θα έχουμε στη διάθεσή μας τις αξιολογήσεις που έχουν ε, γίνει, όταν γίνει η ανάλυση στην οποία σκοπεύω να προβώ των πτυχών στο σύνολό τους του χαρτοφυλλοκίου που θα ε, συζητηθούν στην προσοχή, στις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές. Και αυτό με απόλυτη συνεργασία και διαφάνεια με την Επιτροπή σας. Γιατί? Για να είμαι και τίμια ξέρουν ε, τα μέλη τη Επιτροπής σα πολύ περισσότερα από όσο μπορώ εγώ ποτέ να ελπίζω ότι θα μάθω για το χαρτοφυλάκι αυτό που μου έχει ανατεθεί. Ξέρετε ότι είχα πολύ λίγο χρόνο σε θέσή μου για να ενημερωθώ. Έχετε λοιπόν βαθύτατε γνώσει από ό,τι διαπιστώνω των πτυχών τη πολιτική, ε, του τομέα αυτού πολιτικής ε, και όλων αυτών των θεμάτων. Πρέπει λοιπόν εγώ είμαι υποχρεωμένη να έχω στάση ανοιχτή απέναντί σα και διαφανή και να είμαι έτοιμη να ακούσω τι προτάσει, τι ιδέε σα, το πού θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι, το πώ θα πρέπει να αλλάξει κάτι, εάν θα πρέπει να αλλάξει κάτι και το πώ θα πρέπει εγώ να ανταποκριθώ σε αυτήν την αλλαγή. Παρακαλώ, ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μαρανέσκου. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, λέει ο κύριος Μαρανέσκου. Είμαι πεπισμένος ότι έχετε υπόψη πως υπάρχουν περιορισμοί στην ε, αγορά εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των οποίων πέφτουν θύματα βέβαια και οι ερευνητέ. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προσελκύσει ειδικού επιστήμονε από τρίτε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις γραπτές σας απαντήσεις ε, είπατε πως θα σχεδιάσετε πολιτικές οι οποίες θα προαγάγουν την ελευθερία κυκλοφορίας των ερευνητών και επιστημόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς πολιτικές σκοπεύετε να αναπτύξετε έτσι ώστε να αντιμετωπιστευτεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πέμπτη ελευθερία σημαίνει δημιουργία της ελεύθερης αγοράς της έρευνας ουσιαστικά. Μεταφορά γνώσης, διάδοση της γνώσης που διαθέτουμε. Η ασφάλιση ότι τη γνώση αυτή ε, την ε, εκτιμούμε, την αξιολογούμε στους όρους της όλοι, σημαίνει ταυτόχρονα ότι καταρρύπτουμε τους φραγμούς που αντιμετωπίζει αυτή η πέμπτη ελευθερία. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με το μεστιπλίσμο της δικής μου αρμοδιότητας, απλούστευση φερρυπίν, ταυτόχρονα όμως σημαίνουν και ε, ενθάρρυνση του να επιτύχουμε το στόχο του 3% πάλι στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, ε, επίσης θέματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή ολοκλήρωση επιτέλους του συστήματος του Ευρωπαϊκού ε, διπλώματο ευρεσιτεχνία, αλλά ταυτόχρονα αγγίσουν και τομεί δραστηριοτήτων χαρτοφυλάκια, δηλαδή άλλων επιτρόπων. Και πρέπει να φροντίσουμε, να προσφέρουμε, να αναπτύξουμε και εν τέλει να θεσπίσουμε αυτή την πέμπτη, να θέσουμε σε εφαρμογή, δηλαδή αυτή τη σημαντικότατη πέμπτη ελευθερία. Λίγο πολύ όπω δημιουργήθηκε και η ενιαία αγορά. Ποιοι ήταν οι φραγμοί που αντιμετώπιζε η ενιαία αγορά. Διάφοροι ήταν οι επίτροποι στα χαρτοφυλάκια των οποίων υπήρχε η αντιμετώπιση των φραγμών των εμποδίων η οικοδόμηση ε, γεφυρών. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Όχι μόνο εγώ, αλλά στη συνεργασία και με τους άλλους συναδέλφους επιτρόπους. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τις γέφυρες που χρειάζονται, έτσι ώστε να είναι ουσιαστική η λειτουργία της πέμπτης ελευθερίας, να υπάρξει μια πραγματική εσωτερική αγορά, ενιαία αγορά για την επιστήμη και τη γνώση. Κύριε συνάδελφε, κύριε Μαρινέσκου, συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως θα πρέπει να ε, βεβαιωθούμε ότι θα αξιοποιούνται αποτελεσματικά τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά χρήματα, τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Φορολογού που δαπανώνται για την υπόθεση αυτή. Ποια είναι η θέση σας ως προς την ε, χρηματοδότηση υπό τον όρο ενός ενδεχόμενου ή προσδοκόμενου αποτελέσματος. Ίσως είναι πιο εύκολο να συζητά κανείς ένα τέτοιο ζήτημα παρά να το υλοποιήσει ως ιδέα εν τέλει. Όμως η έρευνα, έρευνα που θα φέρνει αποτέλεσμα, είναι πολύ σημαντική. Και εάν δεν εξασφαλίσουμε αποτελέσματα από την έρευνα, αποτελέσματα τα οποία θα στηρίξουν, θα, βοηθήσουν την οικονομία μας, που θα τις επιτρέψουν να ξεφύγει από την κρίση που διέρχεται τώρα, ε, θα υποβαθμιστεί η έρευνα. Και εγώ δεν σκοπεύω να επιτρέψω κάτι τέτοιο. Γιατί η έρευνα, ο επιστήμονας, μας δίνει εργαλεία και αν χρησιμοποιήσουμε σωστά τα εργαλεία αυτά, σωστά, καλά, μπορούμε να, να έχουμε την καινοτομία, να δημιουργούμε νέες θέσει εργασία. Και είναι σημαντικό πολύ να υποστηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριο Περίλου, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, υποψήφια κυρία Επίτροπε, το πρόγραμμα έρευνα για την έρευνα, το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη τη τεχνολογία είναι ένα κεντρικό εργαλείο τη στρατηγική Λισαβόνα για να δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πιο ανταγωνιστική οικονομία η οποία να βασίζεται στην γνώση. Τα αποτελέσματα που έχουν κτηθεί από τα διάφορα προγράμματα είναι σημαντικά και με τον τρόπο αυτό έχει ευνοηθεί και η συνεργατική έρευνα που εμπλέκει πολλές χώρες. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής τώρα είναι πολύ επίκαιρο και αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στην Κομισιόν στο να δώσει περισσότερα κίνητρα για την έρευνα στη γεωργία. Είπατε θα μπορεί να είναι το ίδιο έτοιμά σας ε, και για κάποια σημαντικά γεωρικά προϊόντα για τα οποία η επιστημονική κοινότητα είναι πεπισμένη ότι περιέχουν ε, θεραπευτικές ουσίες που περιέχονται. Τέτοιες προτάσεις θα πρέπει ήδη να ενταχθούν στα προγράμματα εργασίας του γεωργικού τομέα του 7ου προγράμματος πλαισίου ή στην προετοιμασία ε, του 8ου προγράμματος ε, πλαισίου. Τι άποψη έχετε γι' αυτό. Απάντηση. Η αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος και αρκετά αρκετή έρευνα γίνεται στον τομέα των κλιματολογικών αλλαγών, διότι περίπου μισός από τον προπολογισμό του προγράμματος πλαισίου υποστηρίζει έρευνα που ασχολείται με βιώσιμη ανάπτυξη και ένας από τους βασικούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης βέβαια είναι η καταπολέμηση της κλιματολογικής, των κλιματολογικών αλλαγών. Η έρευνα που χρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται της αναπτύξεως μοντέλων για την αλλαγή του κλίματος και για τη συλλογή στοιχείων που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα και να προβλέψουμε την αλλαγή του κλίματος και τι συνέπειες θα έχουν οι αλλαγές στο οικοσύστημα. Αυτό που αναφέρεται εν ολίγης για τη γεωργία και τι συνέπειες έχει για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και πρέπει να κάνουμε. Και υπάρχουν διάφορα προγράμματα, αρκετά πολλά προγράμματα ερευνητικά, τα οποία ε, αφορούν τον τομέα το γεωργικό τι διαφορά κάνει, παραδείγματο χάρη, αν έχουμε δύο βαθμούς πιο ζεστό κλίμα για προϊόντα ή σοδιές που καλλιεργούνται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Ευρώπης. Οι συνέπειες είναι διαφορετικές για την Νότια Ισπανία από άλλη περιοχή. Οι δύο βαθμοί διαφορά έχουν ανάλογα με το που βρίσκεσαι διαφορετικές επιπτώσεις. Έχουμε καλά χρηματοδοτούμενη έρευνα που ε, ανοίγει το δρόμο προς το μέλλον όσον αφορά αυτούς τους τομείς για να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Και αυτή η έρευνα είναι κρίσιμη σημασίας, είναι πολύ σημαντική και μπορεί να, μπορεί να επηρεάσει και να επηρεάσει αυτό που σας ενδιαφέρει, κυρίως την γεωργία. Έχουμε το πρόγραμμα που προανέφερα, τις πρωτοβουλίες της κοινέ που συναθρίζουν τις δραστηριότητες των κρατών μελών και είναι εξίσου σημαντικέ και μία από τι προτεραιότητε που έχουν επιλεγεί για, το, την πρώτη κοινή πρωτοβουλία αφορά τι συνέπειε τη γεωργία στι κλιματολογικέ αλλαγέ. αυτό είναι ένα παράδειγμα των όσων συμβαίνουν. Θέλετε να κάνετε και συμπληρωματική ερώτηση, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Η έρευνα αφορά διάφορους ε, τομείς τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές, υγεία, περιβάλλον κλπ. Σκεφτήκατε ήδη πώς να συντονίσετε τις ερευνητικές δράσεις των διαφόρων γενικών διευθύνσεων, ούτω ώστε να επιτευθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Εάν σκέφτεται να κάνετε πιο ευέλικτη την διοικητική διαδικασία του 8ου προγράμματος πλαισίου για να διευκολύνετε τον, τη συμμετοχή σε αυτό το πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ. Απάντηση. Ο συντονισμός ερευνητικών δράσεων. Συντονισμός γενικών διευθύνσεων. Η ίδια Γενική Διεύθυνση Έρευνας ε, διεξάγει πάρα πολλές έρευνες που αφορούν άλλους τομείς πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά επί συντονισμένης βάσης, ε, βάση συνεργασίας γίνεται αυτό με αποδοτικότητα και πρέπει να συνεχιστεί όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο το 8ο. Το πρώτο που θα πρέπει να εξετάσω, αν τελικά εγκριθεί ο διορισμός μου, είναι ενδιάμεση εξολόγηση του 7ου προγράμματος ε, πλαισίου Είμαι σίγουρη ότι στην αξιολόγηση αυτή θα συμπεριληφθούν πολλέ προτάσει όσον αφορά τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι αυτό φαίνεται να είναι ένα τομέα που δεν αφορά μόνο αυτή την Επιτροπή, αλλά και άλλου εκτό αυτή τη Επιτροπή. Πολλοί συζητούσαν την έλλειψη συμμετοχή, πώ χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή και τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει κλπ. Και είπα προηγουμένω κάτι που επαναλαμβάνω τώρα. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να εστιαστούμε σε Τομεί που ενδιαφέρουν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να καθορίζουμε τα διάφορα προγράμματα και ζητάμε έρευνα, θα πρέπει να μιλήσουμε με του ενδιαφερομένου, να δούμε τι έχουν να πούν. Κατά κάποιο τρόπο, αν μπορούμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μέσο χρηματοδοτήσεως και μερισμού του κινδύνου για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα βοηθά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που χρησιμοποιούν τεχνολογία εχμή, Να μπορούμε να βοηθήσουμε και τι πιο απλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει και γενικά να καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Next. Ευχαριστώ. Η κυρία Κουτιέρε Κορτίνε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε ε, υποψήφια επίτροπε. <clears throat> Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικά υποστηρίζουμε την Κομισιά. Πολύ περισσότερο από ότι το Συμβούλιο. Βλέπουμε όμως ότι πρόσφατα σε όλες τις γενικές διευθύνσεις υπάρχει μια προσπάθεια των κρατών μερών για την επανεθνικοποίηση του προϋπολογισμού. Αυτό περιλαμβάνει και την εθνικοποίηση του εβδόμου ου προγραμμάτος πλαίσιο. Εδώ αυτό με απασχολεί πάρα πολύ γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει απώλεια ποιότητος και απώλεια δυνατότητας της Ευρώπης να λαμβάνει αποφάσεις με το παλιό άρθρο 169 που δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον. Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση του Κοινοβουλίου <clears throat> για το πώς λειτουργούν αυτά τα προγράμματα, ούτε για το τι χρήματα δίνουν τα κράτη-μέλη και αν επαναθνικοποιούνται αυτά τα ταμεία. Εσείς είσαστε διατεθειμένοι λοιπόν να υποστηρίξετε τον προπολογισμό του 7ου προγράμματος πλαισίου, γιατί είναι η Κομισιόν η οποία πρέπει να αποφασίσει για την κατανομή των προγραμμάτων μέσα στο πλαίσιο αυτό. Θέλετε λοιπόν να το κάνετε αυτό για να διατηρήσετε τα κριτήρια αριστείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κουτιέρας Κορτίνες. Τα πλαίσια, τα προγράμματα πλαίσιο στην Κομισιόν παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι αν εξετάσει κανείς την πολυμορφία της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο εμεί έχουμε χάσει πολλές ευκαιρίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι ανταγωνιστών μας, όπως είπαμε προηγουμένως, η Ινδία, Κίνα, Ηνωμένε Πολιτείες κτλ. Έναντι των άλλων παικτών στην αγορά έρευνα. Εγώ δεν θα ήθελα να επανέλθουμε στο προηγούμενο μοντέλο που χαρακτηρίζεται από έλλειψη συντονισμού και αν δείτε παραγωγικά το δίκτυο αυτό για την ασφάλεια των τροφίμων στο Euronet όπου φάνηκε ότι υπήρχαν 72 χωριστές έρευνες από τα 27 κράτη-μέλη για το ίδιο βακτηρίδιο της σαλμονέλας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα χαμένων απολεσθέντων ελευθεριών όπου η Ευρώπη απέτυχε να λειτουργήσει σαν ενιαίος φορέας και όχι σαν αριθμητικό άθροισμα 27 χωρών. Εγώ δεν θα ήθελα να επανέλθουμε λοιπόν στην επανεθνικοποίηση της έρευνας, όπως λέτε. Αλλά ξέρω ότι θα υπάρχουν πιέσεις από τα κράτη-μέλη και πίεση και μέσα στα κράτη-μέλη για να μειωθούν οι ερευνητικοί προϋπολογισμοί <clears throat> και αυτό θα ήταν πραγματικά μια υπαναχώρηση. Εγώ σίγουρα θα υποστηρίξω τον προϋπολογισμό του προγράμματος πλαισίου 7 μέσα στην Κομισιόν, εάν είμαι αρκετά τυχερή να με εγκρίνεται ως Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Α, συμπληρωματικό ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, εγώ θέτω το ερώτημα αν είσαστε έτοιμοι να μας εξηγήσετε πώς θα λειτουργήσει το άρθρο 175, πώς θα γίνεται ο έλεγχος του προϋπολισμού και ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις για τα κοινά προγράμματα και πώς θα λειτουργήσουν τα προγράμματα αυτά, πώς θα συντονιστούν αυτά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, γιατί αυτό είναι ένας δεύτερος χώρος έρευνας που ελέγχεται από τα κράτη-μέλη. Και τονίζω ότι το Κοινοβούλιο απαιτεί να υπάρχει μια ελάχιστη διαφάνεια για τα θέματα αυτά. Δεν υπάρχει λοιπόν η ίδια διαφάνεια που υπάρχει στο Κοινοβούλιο έναντι της Κομισιόν από την Κομισιόν έναντι του Κοινοβουλίου. Καμία. Κοιτάξτε κύριε Αγκουτιέρες, μεταξύ μας αυτό είναι πραγματική συνεργασία και αν θέλουμε να λειτουργήσει και αν θα πρέπει να υπερασπιστούμε την έρευνα, αν θέλουμε να πετύχουμε πράγματα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, χρειάζομαι την πραγματική υποστήριξή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η υποστήριξή σας. Ανεξάρτητα του έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εκπροσωπείτε και τα 27 κράτη-μέλη και ξέρετε τι συμβαίνει σε κάθε κράτος. Θα πρέπει μαζί να κινηθούμε να καταλήξουμε σε κάποιες αποφάσεις όσον αφορά το μέλλον. Αν θα είναι ευρωπαϊκός ερευνητικός χώρος ή η αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου και τα αποτελέσματα αυτής ή οι συζητήσεις που ξεκινούν για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Για μένα, εσείς είστε εταίροι μου οι μου πρέπει να συμμετάσχετε αν θέλουμε να παραγάγουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα πλαίσιο και τον καλύτερο δυνατόν ευρωπαϊκό ανοιχτό χώρο έρευνα στο μέλλον. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος Τόμψον. Συνάδελφο Τόμψον έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε, θα ήθελα να επιστρέψω στο ερώτημα που αφορά τις γυναίκες και την επιστήμη. Είπατε προηγουμένως ότι θα πρέπει να έχουμε πιο πολλές γυναίκες που θα ενδιαφερθούν για τις επιστήμες. Αλλά στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου συνέταξε έκθεση για τις γυναίκες και τις επιστήμες που δείχνει ότι σήμερα πάνω από 60% των φοιτητών στα πανεπιστήμια είναι γυναίκες, αλλά μόνο 30% των ερευνητών στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Και όσον αφορά τις ανώτατες θέσεις στα πανεπιστήμια, τα στοιχεία είναι πολύ πιο χαμηλά. Σε όλη την Ευρώπη, κατά την άποψή μου, δεν μπορούμε να ανεχθούμε, να μην χρησιμοποιήσουμε τόσο μεγάλο δυναμικό της Ευρώπης, ταλέντο, σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ήδη στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο υπήρχαν κάποια μέτρα για να αυξηθεί ο ρυθμός των γυναικών ερευνητριών που θα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα. Αυτό δεν ισχύει όμως το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και τώρα καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση. Μόλις 20% των χρημάτων για τα ερευνητικά προγράμματα πηγαίνει στις γυναίκες και αυτό δεν συμφωνεί με τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων. Το ερώτημά μου λοιπόν για σας είναι θα βελτιώσετε την ισότητα των φύλων εντός τη Ευρωπαϊκή Έρευνα, εξασφαλίζοντα ότι περισσότερε γυναίκε θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση σύντομη. Η πρώτη είναι ναι. Δεύτερον, η κατάσταση που σωστά περιγράψατε έτσι έχει και είναι απαράδεκτη, όπως αναφέρετε και στην έκθεσή σας. Δεν είναι μόνο θέμα ισότητας, είναι και θέμα σπατάλης ανθρωπίνων πόρων και ταλέντων. Κατά πρώτον, αν επικυρωθεί ο διορισμός μου, θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Γενικέ Διευθύνσει για την έρευνα να αγηθούν. Να δώσω το παράδειγμα. Θα πρέπει να πετύχουμε το στόχο του 40% συμμετοχή των γυναικών σε ομάδε εμπειρογνωμόνων και σε προσπάθειε αξιολογήσεω. Δεύτερον, εάν επικυρωθεί ο διορισμό μου, θα ήθελα να γίνει εξορθολογισμός διαχείριση των διαφόρων ερευνητικών ιδρυμάτων. Θα πρέπει να είναι σωστή διαχείριση και των δύο φύλων. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τι ιδιαίτερε ανάγκε των γυναικών σε φάση συνθήκε εργασία και το καθεστώ των γυναικών. Και ξέρετε, προ καιρού αναφερθήκαμε στη διαφορά αμοιβών. Ήταν μια καινοτομία αυτή ε, που συζητήθηκε η διαφορά αμοιβών μεταξύ των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά θα πρέπει να έχουμε ευαισθητοποίηση και επικοινωνία μια εκστρατεία όπως τότε που κάναμε τη διαφορά των αμοιβών. Θα πρέπει να γίνει εκστρατεία ενημέρωσης που θα εστιάζεται στις νέες κοπέλες ε, από δημοτικό, γυμνάσιο, τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το χώρο εργασίας. Να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες που θα καλύπτουν τις ανάγκες των γυναικών και να μιλήσω με εκείνους εκεί τους τομείς που ήταν επιτυχέστατοι όσον αφορά το να κρατούν τις γυναίκες τους τομείς τους ενώ άλλοι δεν ήταν τόσο επιτυχεί. Μπορούμε να μάθουμε από εκείνου που τα κατάφεραν καλύτερα και θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά που θα μάθουμε. Ε, και να τα δώσουμε αυτά τα μαθήματα, να δείξουμε στου άλλου που δεν τα κατάφεραν τόσο τι έκαναν οι άλλοι. Ευχαριστώ. Επερώτηση. Άλλο ένα σχόλιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απάντηση που δώσατε. Και επίση για το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή 400.000 ερευνητέ, Ευρωπαίοι ερευνητέ, ε, απασχολούνται στι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Μεγάλη απώλεια. Εάν πρόκειται λοιπόν να ε, υλοποιήσουμε τους στόχους Λισαβόνας, χρειαζόμαστε 700.000 ερευνητέ στην Ευρώπη, βάσει τα στοιχεία τη Ευρώπη. Εάν δηλαδή δεν αξιοποιηθεί το γυναικείο δυναμικό, πάλι θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Απάντηση. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σα. Πρέπει με του στόχου που ορίζουμε να ξέρουμε κιόλα ότι θα φέρουμε αποτέλεσμα. Δεν είναι κάποιοι τυχαίοι στόχοι. Είναι στόχοι συγκεκριμένοι και πρέπει να προσφέρουμε συγκεκριμένα μέσα, συγκεκριμένες πολιτικές για την επιτευξή τους. Πιστεύω και ναι, δεν μπορώ ε, παρά να υπογραμμίσω στο μέγιστο βαθμό την ανάγκη και να ε, ε, επικοινωνήσουμε, να διαδώσουμε την ιδέα ότι χρειαζόμαστε και τις γυναίκες. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα φίλων αλλά θέμα ανάγκης και γνώσεων. Ο κύριος Έλερ. Έχουμε μόλις πάρει την αξιολόγηση του έκτου προγράμματος πλαίσιο από την Κομισιόν. Και είδαμε ότι δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της γραφειοκρατίας και του μεγάλου χρόνου για την υπογραφή των συμβάσεων. Έχετε απαντήσει διπλωματικά σε αυτό το επίπεδο ότι θέλετε να κάνετε κάτι, αλλά βέβαια θα πρέπει να προστατεύσουμε και το χρήμα του φορολογούμενου και την ε, σωστή διαχείριση. Αυτή είναι μια διπλωματική όμως απάντηση. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ε, αναθεώρησης του 7ου προγράμματος πλαισίου και πάλι βλέπουμε ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν λειτουργεί το πρόγραμμα αυτό είναι η γραφειοκρατία και η καθυστέρηση. Θέλω λοιπόν μια συγκεκριμένη ε, απάντηση σε ποιο βαθμό είσαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης και τι απάντηση θα δώσετε σε αυτά τα προβλήματα. Κύριε Γκίγαν Κουίν, δεν πρόκειται να ξανα αλλάξω όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στο πρόγραμμα 7, διότι τα γνωρίζετε αυτά. Στο επόμενο, στο προσεχές μέλλον, εάν εγκριθώ από το Κοινοβούλιο, θα προτείνω μια ε, σύσταση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την απλοποίηση. Θα διερευνήσουμε λοιπόν τις επιλογές μας, νέες αντιλήψεις για τη χρηματοδότηση της ε, χρηματοδότησης, μια μεγαλύτερη χρήση των καταποκοπήν ποσών που ανέφεραν ορισμένοι συνάδελφοι προηγουμένω, συναδελφοί σα κύριε Έλλας, και αυτό το αναγνώρισε και το ελεκτικό συνέδριο και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Εγώ είμαι απόλυτα προσιλωμένη στο να εξασφαλίσουμε την συνέπεια και τη συνεκτικότητα. Γιατί μία από τις συνεχείς επικρίσεις που ακούω είναι ότι ξεκινάει ένα σχέδιο και κάποια στιγμή κατά την εκτέλεση αυτού του σχεδίου αλλάζει κάτι. Και τότε <clears throat> υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να έχετε αυτή την ε, απλοποίηση που ζητάτε, αλλά να υπάρχει και μια συνεκτικότητα γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και μεγαλύτερη απλοποίηση στη χρηματοδότηση. Πέραν αυτή τη ανακοίνωση για την απλοποίηση υπάρχουν και τα άλλα θέματα τα οποία ανέφερα προηγουμένω. Δεν μίλησα για το νέο δημοσιονομικό κανονισμό και τη μεταρρύθμισή του. Αυτό θα αλλάξει, θα βοηθήσει τα πράγματα και η πρόταση για το ανεκτό περιθώριο σφάλματος. Αυτό νομίζω θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι λοιπόν αυτά τα συγκεκριμένα θέματα Αυτά είναι τα θέματα που εγώ θα προωθήσω ως πρώτη προτεραιότητά μου αν με εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό. Συμπληρωματικό ερώτημα. Έχουμε μιλήσει και για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ένα από τα κύρια προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται εκεί πέρα είναι το λεγόμενο time to contract, ο χρόνος υπογραφής συμβάσεων. Αυτό δεν είναι στον έλεγχο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά οφείλεται στη δράση της Κομισιόν. Σε ορισμένα προγράμματα αυτός ο χρόνος μεταξύ της αίτησης και της υπογραφής του συμβολέου ανέρχεται σε ένα μέχρι 1,5 χρόνο. Αυτό είναι αδιανόητο για μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, ακόμα και για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό και για τα ελληνικά ιδρύματα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ποια είναι η άποψη σας γι' αυτό. Ναι, βεβαίως και αποδέχομαι τις επικρίσεις σας στο θέμα αυτό. Ήδη στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ε, σημειώνονται σημαντικές περικοπές ε, ως προς αυτές. Βέβαια μπορεί να μην αρκεί, θα πρέπει να κάνουμε κι άλλα και να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο και καθίσταται, πιστεύω, μια άμεση προτεραιότητα να συνεργαστούμε με την Γενική Διεύθυνση ασφαλώ για να βεβαιωθούμε και ασφαλώ αυτό θα επανέλθει στην ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου προγράμματο πλαισίου του προσεχεί δύο-τρει μήνε. Προτεραιότητα είναι, στόχο είναι, ανάγκη είναι να στηρίξουμε τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει στο, πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σανφρός κ. Πάσκα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι θέλετε να δημιουργήσετε έναν ενίο χώρο έρευνας στην Ευρώπη. Με την πέμπτη ελευθερία. Ελευθερία της κυκλοφορίας της γνώσης. Τις αρμοδιότητες όμως για την πνευματική διοκτησία στον τομέα αυτών την έχουν, τις έχουν τα κράτη-μέλη στα χέρια τους και έχουν πολύ διαφορετική στάση. Πώς θα το καταφέρετε λοιπόν αυτό, αυτό το φράγμα πώς θα τον ε, αντιμετωπίσετε. Απάντηση. Για τα δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας. Ήταν ένα θέμα αμφιλεγόμενο τα τελευταία χρόνια. Νομίζω όμως ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι από τα προβλήματα που μας εμποδίζουν στην πρόοδο μας. Είναι ε, μία από τις τροχοπέδες από τις οποίες πρέπει να, τις πρέπει να απαλλαγούμε. Και βεβαίως εφόσον εγκριθούν ε, όλοι οι υποψήφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει μαζί με τους λοιπούς συναδέλφους να συνεργαστώ, όπως και με τη δική σας Επιτροπή, όπως και με τα κράτη-μέλη, να αναζητήσουμε τον τρόπο Τη αντιμετώπιση των προβλημάτων. πώ θα σηκώσουμε τον πύχη στην υπόθεση αυτή και πώ θα αναγνωριστεί καταρχάς ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, ότι δεν επιτρέπει τη συμμετοχή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ορισμένων ανθρώπων, ερευνητών, επιστημόνων και αυτό να το αντιμετωπίσουμε σε συντονισμένο ε, με συντονισμένο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να με πείτε αφελή που πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά πάντως θα προσπαθήσω. Σε συνεργασία και με τον συνάδελφο ε, Επίτροπο εφόσον εγκριθεί η υποψηφιότητά μας και θα προσπαθήσουμε να προκαλέσουμε ένα δημόσιο διάλογο και να ε, προκαλέσουμε ε, δέσμευση σαφή και ελπίζω ότι θα τα καταφέρω και χάρη στη δική σας υποστήριξη, χάρη στην υποστήριξη των μελών της Επιτροπής σας που βέβαια προέρχονται από όλα τα κράτη-μέλη και που έχουν τις απαραίτητες αυτές πολλές και μεγάλες γνώσεις που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους φραγμούς και τις, ε, τα αδιέξοδα. Συμπληρωματική ερώτηση κύριε συνάδελφε. Πιστεύω και εγώ ότι είναι περίπλοκο το ζήτημα. Αλλά βλέπω ότι είστε διαδεθειμένοι να αποδεθείτε στην προσπάθεια αυτή και έτσι σε συνεργασία και με εμά και με τον ε, συναρμόδιο συνάδελφό σα, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να επιτύχετε, να προσπαθήσετε τουλάχιστον να φτάσετε στο στόχο αυτό. Ένα χρονοδιάγραμμα θα μπορούσατε να μας δώσετε μέχρι πότε θα πρέπει να έχει επιλύθει το πρόβλημα. Απάντηση εάν περνούσε μόνο από το δικό μου χέρι, το δικό σα ενδεχομένω η επιτροπή σα, νομίζω η απάντηση θα ήταν αμέσω. Το ταχύτερο δυνατόν. Αλλά βέβαια ξέρουμε ότι δεν είστε μόνο εσεί και εγώ σε αυτή την υπόθεση παράγοντε ε, καθοριστικοί. Αυτό που μπορώ να σα πω αυτή τη στιγμή είναι ότι, θα δεσμε... ότι δεσμεύομαι να συνεργαστώ στενά με τον συνάδελφο επίτροπο και να επιδιώξω την αποδιάρθρωση αυτού του φραγμού, του εμποδίου, της τροχοπέδης, όπως θέλετε πείτε το, ε, το ταχύτερο δυνατό έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την έμπλοκη, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Όλων αυτών δηλαδή που θεωρούν ότι τα προβλήματα τη πνευματική ιδιοκτησία είναι ο μόνο φραγμό που του εμποδίζει από τη συμμετοχή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Εξαντλήσαμε τι ερωτήσει λίγο νωρίτερα από ό,τι είχαμε προβλέψει. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάνω απ' όλα για την πειθαρχία που επιδείξατε και στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις. Και κλείνοντας, θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στην υποψήφια Επίτροπο να πει μερικά λόγια εάν θέλει να ολοκληρώσει την παρουσίασή της. Όπως ήθιστε άλλωστε. Πέντε λεπτά στον υποψήφιο για να λάβει το λόγο. Κύριε Κινγκούρη, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι προσήγγισα τη σημερινή ακρόαση με εστιασμένο τρόπο. Προσπάθησα να κάνω όσο πιο καλή προετοιμασία μπορούσα και πρέπει να πω έτσι προσωπικά ήταν σαν να, σαν να περνάω τις εξετάσεις απολυτής στο γυμνάσιο στη χώρα μου που το ένιωσα πιο πολύ όταν πέρναγα τι εξετάσει η γη μου από ότι όταν πέρναγα εγώ τι εξετάσει. Πιστεύω, όπω είπα και στην αρχή, ότι ο έλεγχο και ο διάλογο είναι στο επίκεντρο τη ευρωπαϊκή μα δημοκρατία. Διεξήχθη συζήτηση που κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και υπάρχουν και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να είχαμε συζητήσει. Έμαθα ότι έχουμε πολλές κοινέ ανησυχίες, άκουσα προσεκτικά τις ανησυχίες αυτές και για εκείνους που είναι στην πολιτική ζωή όπως εσείς και εγώ η έρευνα, η καινοτομία και η πολιτική για τις επιστήμες τι αφορά. Αφορά το να βρούμε και να εφαρμόζουμε ευφύς λύσεις στα κοινά μας προβλήματα. Άρα χρειάζεται εμβάθυνση, ανάπτυξη ε, των πόρων για να αντιμετωπίσουμε τα πλέον κρίσιμα προβλήματα ε, της Ευρώπης. Θα πρέπει να πετύχουμε οικονομική ανάκαμψη, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κλίματος, θα πρέπει να αναπτύξουμε οικονομία με χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος, θα πρέπει να βρούμε λύσεις για υγιή γύρανση, να ενισχυθεί η διεθνή συνεργασία. Βραχυπρόθεσμα, τι σημαίνει αυτό για όλους μας. Η καινοτομία να ηγείται του σχεδίου ανακάμψεως και να χρησιμοποιήσουμε το όραμά μας για το 2020 για να ξανασυναρμολογήσουμε με φύ τρόπο την οικονομία. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και να προστέψουμε το μέσα των προγραμμάτων πλαισίων, θα πρέπει να είναι πιο προσβάσιμα, όπως είπαν όλοι εδώ, ε, να συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι και να είναι φιλικότερα τα προγράμματα για του χρήστε, κυρίω στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Θα πρέπει να εργαστούμε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να ετοιμάσουμε την ενή αγορά για την καινοτομία. Όπω είπα, χρειάζεται συνεργασία με το Κοινοβούλιο και για μένα ιδιαίτερα συνεργασία χρειάζεται με αυτή την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουμε το πολιτικό μα κεφάλαιο από κοινού για να ολοκληρώσουμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα. Χρειάζεται στενή συνεργασία με τα κρατημέλη σε κοινά προγράμματα και αποτελεσματική διακυβέρνηση και θα πρέπει να κινηθούμε και δημιουργικά με τον ιδιωτικό τομέα και άλλου εταίρου για να κινητοποιήσουμε επενδύσει σε καινοτόμε αγορέ. Εγώ προσβλέπω στην πρόκληση αυτή και ελπίζω ότι θα με εγκρίνει, θα με επικυρώσει στη θέση μου το Κοινοβούλιο διότι έρευνα, καινοτομία και επιστήμε για πρώτη φορά να συναθριστούν και να μπουν στο επίκεντρο πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αυτό είναι κάτι που δίνει τεράστιε δυνατότητε για όλου μα. Ξέρω ότι πέντε πολύ στα σοβαρά τη εργασία σα και εγώ το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται συνεργασία, να συνεργαστούμε ως πολιτικοί, διότι αυτό είμαστε όλοι στην αίθουσα. Είπα ότι αν θέλετε έναν δημόσιο υπάλληλο, έναν τεχνοκράτη, ένα γραφειοκράτη, έχετε λάθο άτομο μπροστά σα. Εγώ είμαι πολιτικό, είμαι άνθρωπο που θέλει να κάνει πράγματα. Θέλω να πετυχαίνω αποτελέσματα. Μπορώ να πετύχω αποτελέσματα μόνο έχω την υποστήριξη όλων στην αίθουσα. Αυτό σημαίνει ότι η καινοτομία είναι ουσιαστικά κάτι που μας αφορά εμάς, δηλαδή να διαχειριστούμε όλοι μαζί τις αλλαγές, να ελέγχουμε τις αλλαγές, αντί να μας ελέγχουν οι αλλαγές. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια οικονομία που από σκέψη οδηγεί σε πράξη. Χρειάζεται συνεργασία μαζί σα και μέσω τη συνεργασία ελπίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πνεύμα ανακάλυψη που το υπήνει στην Ευρώπη. Ένα, μια Ευρώπη που θα είναι πρωτοπόρο για στενότερη ε, συνεργασία στην Ένωση, πιο καινοτόμα Ένωση. Ελπίζω ότι σήμερα είναι η απαρχή αυτού του ενδελεχέστερου διαλόγου και σα εγγυώμαι ότι θα υποστηρίξω ότι μπορώ και θα είμαι ανοιχτή. Ε, θέλω να πω ένα πράγμα σας εγγυώμαι επίσης ότι θα είμαι ανεξάρτητη όσον αφορά τον τρόπο σκέψεώς μου και ξέρω πολύ καλά ότι ήρθα ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής κατά το παρελθόν ε, δύο φορές. Και μετά, όπως και σε αυτή την περίπτωση, αν επικυρωθεί ο διορισμός μου, θα πρέπει να ε, δώσω όρκο ανεξαρτησίας. Όπως και ο κ. Σοντή και οι συνάδελφοί του κατά το παρελθόν, πρέπει να μην αμφισβητείτε εγώ πέρασα σχεδόν 10 χρόνια εργαζόμενη ως ανεξάρτητο μέλος Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου. Ελπίζω ότι σήμερα είναι η αρχή ενός βαθύτερου διαλόγου, συζητήσεως και προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ δύο ομάδων πολιτικών ούτως υπήν και ότι εν τη συνεργασία αυτή θα μπορέσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Αυτό περιμένει ο κόσμος εκεί έξω. Τι θέλει ο κόσμος, θέλουν δουλειές για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους θέλουν ασφαλέστερο, καθαρότερο περιβάλλον, θέλουν ε, χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, θέλουν πράσινη ευφυή τεχνολογία. Αυτά είναι λόγια βέβαια, αλλά τα λόγια αυτά μπορούν να γίνουν πράξη μόνο με πραγματική τελιστική πολιτική. Και να σας πω τελικά ότι ξέρω ότι ήθιστο κατά το παρελθόν μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κοινοβουλίου να περιμένουν οι επίτροποι να προσκληθούν οι άνθρωποι στο κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ζητήσω, κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την περίσταση, εάν όσο αρχίζω να μαθαίνω την ε, πολιτική των δύο γενικών διευθύνσεων για, την οποία, για τις οποίες θα είμαι υπεύθυνη, όπως θα μαθαίνω να μπορέσω να έρχομαι στο κοινοβούλιο, να μην περιμένω πρόσκληση, να μπορώ να έρχομαι στο κοινοβούλιο, να ζητώ να μου πείτε ποιες είναι οι απόψεις σας για τους συγκεκριμένους τομείς ε, πολιτικών, που ήταν και θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομίας και να ε, είναι στο επίκεντρο και να είναι κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Είμαι πολύ ευγνώμων πραγματικά ε, για τις συμπληρωματικές πληροφορίες ε, που έχω συλλέξει σήμερα εδώ και ελπίζω πραγματικά ότι θα είναι καλή συνεργασία μεταξύ μας ούτως ώστε την επόμενη πενταετία ή σε πέντε χρόνια να μπορώ να έρθω εδώ και να πω είμαι υπερήφανη για όλα όσα κάναμε. Όχι μόνο εγώ, αλλά αυτά που κάναμε μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος όλων των συναδέλφων, σας ευχαριστώ θερμά. Μια συζήτηση πολύ, ε, πολύ ζωντανή, για πολύ σαφείς τοποθετήσεις, για την πειθαρχία που επιδείξατε η ΜΕΝ και η ΔΕ στις ερωταποκρίσεις. Ήταν τρεις συναρπαστικές ώρες αυτές που περάσαμε μόλις τώρα και σας εύχομαι καλή δουλειά από εδώ και μπρος, καλές επαφές, κάθε τύχη. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ του συναδέλφου γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη δουλειά μέσα σε τόσο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο συνεχίζουμε.